La conférence de presse, c'était bien Oui. Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε εκ νέου. Έχουμε κάποια λεπτά καθυστέρηση και σας ζητώ συγγνώμη. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τους εκπροσώπους της Όλευ, της Ιντερπόλ, της Europol και της Κόζη. και τώρα θα αφιερωθούμε στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων για το σκοπό της σεξουαλικής ή της εκμετάλλευσης. Αυτό το πάνελ θα μας κάνει να κατανοήσουμε πώς τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή εκατομμυρίων ατόμων στον κόσμο. Η εμπορία ανθρώπων και η εκμετάλλευσή τους για σεξουαλικούς σκοπούς ή για σκοπούς εργασιακής εκμετάλλευσης ήταν αντικείμενο πολλών μελετών με μια εικόνα ιδιαίτερα ζωφερή. Σήμερα θα ακούσουμε τον Ντούκο Βανχίλη, τον εκπρόσωπο της Frontex, που θα μας εξηγήσει καλύτερα αυτό το θέμα από μια ευρωπαϊκή σκοπιά και κατόπιν θα ακούσουμε την κυρία Μπίτ Άντερες ε, από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας που θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης του οργανισμού της ε, κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Και όπως σήμερα το πρωί θα οργανώσουμε τη συζήτησή μας με τον ίδιο τρόπο. Οι εισηγητέ μα θα έχουν στη διάθεσή του 15 λεπτά ο καθένα και σα παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από τον εισηγητή και του συντονιστέ. Δύο λεπτά θα έχετε στη διάθεσή σα και κατόπιν θα ξαναδώσω το λόγο στου προσκεκλημένου μα και αν έχουμε χρόνο θα συνεχίσουμε με τι ερωτήσει. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Ντούκ Βαν από τη Frontex που θα μας παρουσιάσει την δική του σκοπιά, μια ευρωπαϊκή προοπτική. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Τίκο Φανχέιλ, δουλεύω για την Frontex ε, στην Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων και ρόλος μου είναι η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων της Frontex σε σχέση με την καταπολέμηση τις εμπορίας ανθρώπων. Η Επιτροπή σας μου ζήτησε να κάνω μία παρουσίαση για το θέμα αυτό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είμαι εδώ. Θα αρχίσω λοιπόν με αυτές τις διαφάνειες. Δεν ξέρω αν τις βλέπετε καλά. Έτσι καλλιώς στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου υπάρχει η παρουσίασή μου. Οπότε θα βρείτε και εκεί τα στοιχεία. Το 2008 άρχισε Frontex τη συλλογή στοιχείων για την εμπορία ανθρώπων. Συλλέξαμε πολλά στοιχεία από τα κράτη-μέλη και από τις χώρες μέλη του Σέγγεν. 30 μέλη είμαστε στην Frontex γιατί είναι και η Ολλανδία και η Ισλανδία και η Νορβηγία στο Σέγγεν. 27 χώρες λοιπόν έδωσαν στατιστικά δεδομένα. Ανεθνικότητα βασίζονται στη, στα στοιχεία που υπάρχουν για την σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά όχι μόνο και για την καταναγκαστική εργασία. 27 χώρες λοιπόν αυτές το 2009, 7.000 θύματα δήλωσαν ότι εντόπισαν. Ποιος είναι ο ορισμός ε, τώρα του εντοπίστηκαν θύματα, γιατί κάποιοι μπορεί να ζήτησαν βοήθεια, κάποιοι προστασία, Τώρα η Επιτροπή συλλέγει στοιχεία προκειμένου να συλλέξει όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία από τις χώρες μέλη που μερικές φορές δεν είναι συγκρίσιμα. Αλλά για μας τη Frontex πρέπει να τα έχουμε γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα νούμερα. Πάντως τα νούμερα αυτά από όλες αυτές τις χώρες μέλη πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι συγκρίσιμα. Κοιτάξαμε λοιπόν τις διάφορες εθνικότητες. Ε, ασχολούμαστε με τα εξωτερικά σύνορα, έτσι, όχι με το τι γίνεται στο εσωτερικό. Από τις 7.000, τα 2.500 περίπου ήταν στο εσωτερικό. Οι περισσότερες είναι γυναίκες, από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία κυρίως. Για άλλε εθνικότητες δεν είχαμε στοιχεία. Πάντως τα υψηλότερα νούμερα θυμάτων είναι από την Νιγηρία, κυρίως γυναίκες και κυρίως για σεξουαλική εκμετάλλευση. Και πολλά παιδιά μάλιστα, 900 από τις 7.000. Στη συνέχεια έχουμε την Κίνα και τη Βραζιλία, 270 και 200 αντίστοιχα. Αλλά όπως σας είπα πολλές φορές δεν εντοπίζονται τα θύματα παρκώς έτσι. Μετά έχουμε το Μαρόκο. Αυτό ήταν έκπληξη για μας για το 2009, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν 120 ε, θύματα που εντοπίστηκαν από το Μαρόκο. Εμείς σε τέτοια στοιχεία θέλουμε να επικεντρωθούμε, σε κάποιες ε, εθνικότητες που αποτελούν έκπληξη για μας. Τώρα στην Ευρώπη, τι διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε την εμπορία ατόμων. Έχουμε την οδηγία βέβαια, η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Συνεπώς, τα κράτη-μέλη το 2013 πρέπει να την εφαρμόσουν και οι διάφορες υπηρεσίες δραστηριοποιούνται ώστε να προσαρμόσουν το έργο τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδηγίας. Η οδηγία αυτή λοιπόν λέει ότι είναι σοβαρό έγκλημα και βέβαια μεγάλη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο σημαντικό και για τις διάφορες, διάφορους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα κράτη-μέλη κατά πολέμηση του εγκλήματος αυτού. Έχουμε βέβαια την συντονιστική μονάδα για τις διάφορες δραστηριότητες κατά πολέμηση στις εμπορίες ανθρώπων. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλους τους φορείς που ασχολούνται με αυτό το θέμα και να συντονίσουμε τις δραστηριότητες όχι μόνο στις χώρες μέλη μεμονωμένα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή σύντομα τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν όλα έναν αξιωματούχο που να έχει αυτό το συντονιστικό ρόλο. Είχαμε μία μέρα κατά της ε, εμπορίας το 2011, όπου οι διευθυντές των διάφορων υπηρεσιών συναντήθηκαν και υπέγραψαν μία κοινή δήλωση για να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης από κοινού, σε συνεργασία δηλαδή μεταξύ τους, να αυξήσουν τον αριθμό των ερευνών και των διώξεων, να κατάσκουν περιουσιακά στοιχεία, να αυξήσουν τον αριθμό των ομάδων των μεικτών, που ασχολούνται με την δίωξη, όπως η Interpol και η Europol που συνεργάζονται, να αναπτύξουν νέα μεθοδολογία όσον αφορά την εκτίμηση των απειλών και να μοιραστούν καλύτερα τις πληροφορίες που διαθέτουν μεταξύ τους. Αυτό, αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο έγινε πέρυσι. Πριν από δύο εβδομάδες υπήρξε και μια ευρωπαϊκή στρατηγική που δημοσιεύθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάστηκε με συνέντευξη τύπου στις 19 Ιουνίου. Στη στρατηγική αυτή, λοιπόν, υπάρχουν διάφορα πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στην επόμενη πενταετία. Κάποιες προτεραιότητες κλειδί είναι καλύτερος εντοπισμός και προστασία των θυμάτων, αύξηση της δίωξης των ε, εμπόρων αυτών ανθρώπων ανάπτυξη επίσης συστημάτων προστασίας των παιδιών, γιατί τα παιδιά βλέπετε ε, πάντα επιδέχονται ιδιαίτερη προσοχή και στην οδηγία, αλλά και ε, οι διάφοροι οργανισμοί ασχολούνται μαζί τους περισσότερο. Επίσης, θέλουμε και μονάδες που εφαρμόζουν τον νόμο σε εθνικό επίπεδο και που συνεργάζονται μεταξύ τους. Και θέλουμε επίσης και μικτές ερευνητικές ομάδες όπου συμμετέχουν και εθνικές αρχές αλλά και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Έχουμε λοιπόν τη δήλωση, έχουμε την ε, οδηγία, έχουμε το συντονισμό. Όλα αυτά αποτελούν εργαλεία μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι διάφοροι οργανισμοί για να πετύχουν τον κοινό στόχο και να δουλέψουν έτσι συντονισμένα. Η εμπορία ανθρώπων είναι, όπως είπαμε, έγκλημα και λαμβάνει χώρα με διαφορετικούς τρόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπόλ ίσως βέβαια να το έχετε ακούσει αυτό και το πρωί, έχει ένα πρόγραμμα με την COSI που ονομάζεται Impact THB, για την αντιμετώπιση δηλαδή της εμπορίας ανθρώπων. Εδώ συμμετέχουν πέντε οργανισμοί και χώρες μέλη, προκειμένου να πετύχουν στρατηγική σημασίας στόχους. Έχουν προτείνει δράσεις που επικεντρώνονται σε 8 στρατηγικούς στόχους. Βέβαια υπάρχει και κάποια επικάλυψη, γιατί όπως είπαμε υπάρχει η στρατηγική, αλλά υπάρχει και οδηγία. Υπάρχουν και τόσα συμφώνησαν οι διευθυντές των οργανισμών μεταξύ τους. Βλέπετε δηλαδή εδώ ότι υπάρχει συνεργασία πάνω στα ίδια θέματα, προκειμένου να ακολουθήσουμε μια κοινή προσέγγιση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τη νέα στρατηγική και για το πρόγραμμα αυτό είναι ότι ζητάμε από τα κράτη-μέλη να έχουν στη διάθεσή τους μηχανισμούς ώστε να ξέρουμε άπαξ και εντοπιστεί ένα θύμα τι πρέπει να κάνουμε με το άτομο αυτό, τι πρέπει να κάνουμε με τις πληροφορίες που έχουμε γύρω από την περίπτωσή του. Οπότε, Θέλω να σας πω λιγάκι τι κάνουμε εμείς συγκεκριμένα με τους 4.000 συνοροφύλακες που έχουμε αναπτύξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα σύνορά της. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στον εντοπισμό και μετά θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Ορισμένοι συνεροφυλάκε έχουν ερευνητικέ αρμοδιότητε. Δεν θέλω όμω να επικεντρωθώ πάνω σε αυτό, γιατί αυτό είναι ρόλο κυρίω τη Europol. Εγώ θα επικεντρωθώ στο τι κάνουμε ε, μαζί με τους συνοριοφύλακες και πώς με τι δράσεις προσπαθούμε να προλάβουμε τα εγκλήματα αυτά. Έχουμε αναπτύξει ένα εγχειρίδιο κατάρτισης βάσει του οποίου γίνεται συνειδητοποίηση. Θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Έτσι, ώστε οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν και να έχουν τα ίδια στοιχεία στη διάθεσή τους τα βάση μυστικών υπηρεσιών έχουμε αναπτύξει και ένα άλλο εγχειρίδιο το οποίο είναι χρήσιμο για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργούν οι εγκληματικές οργανώσεις. Έχουμε επιλέξει τις πρώτες πέντε εθνικότητες, τώρα έχουμε φτάσει στις 7, οπότε εξηγούμε εδώ ποιο είναι το modus operandi, πώς δηλαδή πρέπει να λειτουργούν οι συνοροφύλακες έτσι ώστε να μπορούν να συλλάβουν τους υπεύθυνους. Επίσης υπάρχει και ένα εγχειρίδιο για τον εντοπισμό και την δίωξη των εγκληματικών οργανώσεων που ασχολούνται είτε με την εμπορία ατόμων είτε με το λαθρεμπόριο και ε, στα ε, σύνορα στα αεροδρόμια. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της ε, Aeropol το Impact. Στηρίζουμε το πρόγραμμα SEPOL που είναι και αυτό πρόγραμμα κατάρτισης. Φέτος τα προγράμματα κατάρτισης έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την εμπορία ατόμων. Ε, πρόσφατα πήγαμε και στην Κίνα προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τους εκεί συνοριοφύλακες βάσει του νέου μας εγχειριδίου για το θέμα αυτό. Ε, είδαμε, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε για να οργανώσουν και αυτοί κέντρα υποδοχής ε, ατόμων από άλλες χώρες. Και έτσι ελπίζω κάποια στιγμή ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε πιο αποδομητικά ε, μαζί τους και πιο αποτελεσματικά. Επίσης, στηρίζουμε και διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι τα στοιχεία που δίνει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ή τα στοιχεία που σας έδωσα εγώ, σίγουρα είναι πολύ πιο χαμηλά και ιδίω τα δικά μα σίγουρα είναι πολύ πιο κάτω από τα στοιχεία που θα σα δώσει το Διεθνέ Γραφείο Εργασία. Αυτό το δείχνει, δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα είναι ο εντοπισμό των θυμάτων. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνδυτοποίηση και στους νεροφύλακες και στην αστυνομία, αλλά όχι μόνο, και στους δικαστές, τους ανακριτές, στα νοσοκομεία, μεταξύ των γιατρών, να υπάρξει συνδυτοποίηση, ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων και έτσι σιγά σιγά να μπορέσουμε να έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία για τα θύματα, να φτάσουμε πιο κοντά στα στοιχεία που δίνει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να βγει από αυτό το δράμα που ζει ως θύμα. Αυτά είχα να πω προς το παρόν, αυτή ήταν η παρουσία μου, νομίζω ότι τήρησα το χρόνο μου και έτσι ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σεβαστήκατε απόλυτα το χρόνο και σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Άντρες, η οποία θα μας ε, παρουσιάσει το πρόγραμμα δράσης ε, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Παρακαλώ. Thank you, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ, Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω όλους. Ο, οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας συνήθως δεν είναι εμπειρογνώμονος για θέματα εγκληματικότητας, κυρίως για θέματα εργασίας. Αλλά βεβαίως ε, εντοπίσαμε την εργασία μας στον τομέα αυτό και πριν σας παρουσιάσω τα νούμερα, τους αριθμούς, τα στοιχεία τα οποία ο κύριος ε, Μαρτίβε μόλις σας ε, περιέγραψε, θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω κάποια στοιχεία όσον αφορά την ε, καταναγκαστική εργασία. Ξέρετε ότι υπάρχει ο ορισμός βάσει του πρωτοκόλλου του Παλέρμο για την εμπορία ανθρώπινων όντων και η καταναγκαστική εργασία είναι ένας από τους σκοπούς και τις αιτίες που υπάρχει αυτή η εμπορία ανθρώπινων όντων. Όσον αφορά λοιπόν τον ορισμό αυτής της καταναγκαστικής εργασίας, βασίζουμε εδώ στη Σύμβαση 29, 1930, πρόκειται ουσιαστικά για την αρχαιότερη σύμβασή μας. Πρόκειται λοιπόν για μια εργασία η οποία ασκείται υπό απειλή και χωρίς οικειοθελώς ε, το ίδιο το άτομο να προσφέρει την υπηρεσία ή την εργασία αυτή. Κοιτώντα λοιπόν αυτόν τον ορισμό, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει άμεση σχέση με την εμπορία ανθρώπων, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο του Παλέρμο, και βεβαίως καλύπτει όλες τις πτυχές αυτής της εμπορίας ανθρώπινων όντων και δεν συμπεριλαμβάνεται στη δική μας ανάλυση η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εμπορία οργάνων. Εντοπίζουμε λοιπόν την προσοχή μας στην καταναγκαστική εργασία και την σεξουαλική εκμετάλλευση. Το πρόγραμμα του οργανισμού μας επεκτείνεται σε πάνω από 40 διαφορετικές χώρες και θα δείτε στα νούμερα που θα σας παρουσιάσω ότι αυτό δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή υπάρχει η αλυσίδα προσφράση και ζήτησης, έχουμε σήμερα πολλούς ε, αριθμούς και στοιχεία που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιους τομείς, παραδείγματο χάρη, όπως την κλωστοδιφαντουργία, όπως ε, την αλληλεία, τα είδη διατροφής, τη γεωργία και Γι' αυτό και εντοπίζουμε κάποια από τα στοιχεία μας, ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία τα οποία εχθές ανακοινώθηκαν ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι 20,9 εκατομμύρια ανδρών, γυναικών και παιδιών που είναι θύματα αναγκαστικής εργασίας. Και όπως βλέπετε εδώ από αυτήν την διαφάνεια, οι περισσότεροι οι οποίοι είναι θύματα αυτής της εκμετάλλευσης στον τομέα της γεωργίας, τη κατασκευαστικό τομέα, ε, οικιακή εργασία, 22% είναι και σεξουαλικά εκμεταλλευόμενοι και οι υπόλοιποι είναι θύματα αυτής της εκμετάλλευσης από στρατιωτικό ε, δυνάμεις, ε, στις ε, φυλακές. Βλέπετε εδώ την κατανομή την γεωγραφική. Η μεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται στην Ασία και τον Ειρηνικό. Βλέπετε εδώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που σε σχέση με τις άλλες αναπτυγμένες περιοχές, δηλαδή την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία, 1,5 εκατομμύρια θύματα για τον αναπτυγμένο χώρο. Για την Ανατολική Νότια Ευρώπη 1,6 εκατομμύρια είναι τα θύματα. Αν κοιτάξουμε εδώ τις επικρατέστερες τάσεις, γιατί αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό για να κατανοήσει κανείς την κατανομή στις γεωγραφικές περιοχές. Βλέπετε την ε, Νοτιοανατολική Ευρώπη και χώρες της πρώην ε, Σοβιετικής Ένωσης, της Κοινοπολιτείας 4,2 εκατομμύρια, συγγνώμη, 4,2 της χιλής στις αναπτυγμένες ε, οικονομίες 1,5 είναι αυτό το ποσοστό. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε την κατανομή αναφύλου. Άνδρες, γυναίκες και εδώ βλέπετε, βέβαια δεν εκπλήσει αυτό κανένα, την στη σεξουαλική εκμετάλλευση η μεγάλη πλειοψηφία, 98% είναι γυναίκες, κορίτσια. Στην καταναγκαστική εργασία οικονομική εκμετάλλευση η πλειοψηφία είναι άνδρες. 55% συνολικά πάντως είναι γυναίκες, συνολικά και 45% ε, ο ανδρικός πληθυσμός. Κοιτάξαμε επίσης και την σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτής της εκμετάλλευσης και της κινητικότητας της μετανάστευσης και στο εσωτερικό μιας χώρας αλλά και εκτός. Και υπάρχει μια σαφή σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης η πλειοψηφία των θυμάτων που τελικά έγιναν σεξουαλικά θύματα είναι μετανάστες τις πιο πολλές φορές εκτός της χώρας τους. Βρήκαμε λοιπόν και κάποια στοιχεία που προέρχονται από τις διοκτικές αρχές και είδαμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες που αναγκάζονται να υποστούν αυτή τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η πλειοψηφία λοιπόν είναι γυναίκες. Η πλειοψηφία των θυμάτων δεν αναγκάζονται να βγουν εκτός της χώρας τους. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι τα πιο πολλά θύματα βγαίνουν και εκτός της χώρας τους, αναγκάζονται δηλαδή να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, αλλά και πολλές φορές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χτεσινή παρουσίαση που κάναμε, πιο συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδατε τους συνολικούς αριθμούς. Εδώ είναι η εικόνα μόνο των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 380.000 είναι ο συνολικός αριθμός και εδώ είμαστε πολύ συντηρητικοί αλλά δεν μπορούμε αξιόπιστα να ανακοινώσουμε κάτι άλλο. Η πλειοψηφία είναι γυναίκες, 58% αυτών είναι γυναίκες και οι επικρατέστερες τάσεις, όπως βλέπετε εδώ, 1,8 θύματα της χιλής. Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας σε σχέση με την σεξουαλική εκμετάλλευση. Αν κοιτάξουμε τώρα, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία των διοκτικών αρχών, τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά αυτό βεβαίως έχει άμεση σχέση αυτό που μόλις σας είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ότι δηλαδή υπάρχει θέμα εντοπισμού όταν ε, οι αρχές των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συλλέγουν στοιχεία για άλλες αγορές από αυτήν τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δεν μπορούμε δυστυχώς να μπούμε περισσότερο στα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για να καταλάβετε πώς φτάσαμε στην προβολή αυτών των στοιχείων και σε αυτά τα συμπεράσματα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στηριχτήκαμε σε όλες τις πιθανές ε, πηγές στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε, εντοπίζοντας κυρίως πηγές ε, από πολλές χώρες, διαφορετικές γλώσσες, με τις δύο ομάδες εμπειρογνωμόνων που είχαμε για το θέμα αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις για το θέμα αυτό, αλλά αυτό εξηγεί κατά κάποιο τρόπο τα διαφορετικά στοιχεία που δίνουμε εμείς σε σχέση με τα στοιχεία ε, των άλλων πηγών. Θελήσαμε να έχουμε μία πιο ε, ολοκληρωμένη εικόνα από αυτή που έχουν οι διοκτικές αρχές και γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορές στα στατιστικά στοιχεία. Στην βάση δεδομένων έχουμε πάνω από 8.000 περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας. Κοιτήξαμε ποιες είναι, είναι τα χαρακτηριστικά των θυμάτων. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κοιτώντας ε, την πλειοψηφία των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την καταναγκαστική εργασία, τα περισσότερα θύματα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βεβαίως και άτομα που προέρχονται από την Ασία, την Αφρική και την χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά η πλειοψηφία αυτών των θυμάτων είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τομείς στους οποίους εργάζονται είναι η γεωργία, κατασκευαστικός τομέας, βιομηχανικός και οικιακή εργασία και ο κύριος ε, τρόπος καταναγκασμού είναι η κράτηση των ε, διαβατηρίων και εγγράφων ταυτότητας, καθώς και η κράτηση των μισθών τους. Και βεβαίως ε, αυτά τα δύο γεγονότα περιορίζουν τη δυνατότητα κυκλοφορίας. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα περισσότερα από αυτά τα θύματα ζούσαν σε πάρα πολύ δύσκολες ε, συνθήκες. Αυτό βεβαίως δεν είναι, ε, αν θέλετε, το μόνο ενδεικτικό στοιχείο για την καταναγκαστική εργασία, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη. Η μελέτη μας έδειξε βεβαίως ότι υπάρχουν και τα στοιχεία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ διαπιστώσαμε κάτι που το είχαμε δει και από τη δική μας έρευνα, ότι η ζητιανία είναι, στα παιδιά είναι επίσης ένας τρόπος εκμετάλλευσης των παιδιών και αυτό γίνεται πολύ συχνά από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. Όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, θα σας κάνω κάποια σχόλια καθότι όπως σας είπα προσπαθήσαμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των εγκληματιών αλλά και των θυμάτων. Σήμερα η δίωξη, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιο αυστηρή όχι βέβαια όσο αυστηρή θα θέλαμε, για τα θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, για τους ε, εγκληματίες ε, που εκμεταλλεύονται σεξουαλικά Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι θύτες και τα θύματα ανήκουν στην ίδια εθνικότητα αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει πάντα σε όλο το, τις περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, της οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως παραδείγματο χάρη της ε, φοροδιαφυγής. Και επαναλαμβάνω ότι κάτι που ήδη το ξέραμε μπορέσαμε να το αποδείξουμε και με τα στοιχεία, ότι δηλαδή υπάρχει συχνά η ίδια ε, ε, εθνικότητα μεταξύ των θητών και των θυμάτων και πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς μία νόμιμη από μία ημινόμιμη ή εγκληματική δραστηριότητα. Πολλές φορές στη διαχωριστική γραμμή είναι πολύ δύσκολο να τεθεί. Νομίζω ότι δεν έχω άλλο χρόνο, θα σταματήσω λοιπόν, αλλά όπως σας είπα όλα αυτά τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί καθώς και η μέθοδος εργασία μας και το πλαίσιο στο οποίο εργαστήκαμε. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και να βρείτε την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ο κύριος Νιτοντάν για τους φιλελευθέρους για δύο λεπτά. Ξεκινάμε τους συντόνιστές λοιπόν. Ευχαριστώ και τους ε, δύο μιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ε, καταρχήν να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Frontex. Ε, ποια είναι η διαδρομή από την Ιγυρία. Θα ήταν ενδιαφέρον να το γνωρίσουμε αυτό και αναφέρατε ένα συντονιστή, ε, μία συντονίστρια μάλλον, αναφερθήκατε σε μία γυναίκα που είναι αρμόδια για το συντονισμό της της εμπορίας ανθρώπων. Ποιο είναι αυτό το άτομο. Επίσης, ε, αναφερθήκατε σε 400 Βέλγους συνοριοφύλακες. Ε, δεν έχει νόημα για μένα αυτό εννοούσατε. Ίσως να μην άκουσα καλά τέταρτον. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια αντίγραφα του εγχειριδίου. Είπατε ότι εκπονήσατε ένα εγχειριδίο για να δείξετε πώ λειτουργούν αυτέ οι συμμορίε. Θα ήταν κάτι πολύτιμο για μα. Πέμπτον, μπορείτε να μα δώσετε κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε για την Κίνα και την κατάρτιση των Κινέζων συνοριοφυλάκων. Ε, γιατί είναι πολύ ενθαρρυντικό αν οι Κινέζοι ε, αρχίζουν τώρα να συμμετέχουν στην καταπολέμηση του προβλήματο. Και τέλο, τι θα έπρεπε να κάνει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα πρέπει να συστήσει η Επιτροπή μας που θα βοηθούσε το έργο σας. Ε, ποια μέτρα θέλετε να εισαγάγει η Ένωση στην εκπρόσωπο του ΔΟΕ. Μια ερώτηση. Αναφερθήκατε στους ορισμούς και να ρωτήσω αν σας κατάλαβα καλά. Αναφερθήκατε σε θύματα που δεν ε, είχαν ε, πάει εκούσια, αλλά από ό,τι κατάλαβα τα περισσότερα θύματα αρχικά πάνε εκούσια, δηλαδή του λένε θα έχετε μια καλή δουλειά, θα περάσετε καλά, δώσουμε το διαβατήριό σου και θα περάσουμε πολύ ωραία. Ίσως ε, το θέμα είναι να το ορίσουμε πότε ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για κάτι τρομερό και όχι για ευχαρίστηση. Και επίση, τι θα πρέπει να συστήσει η Επιτροπή μας τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει τα πράγματα, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Νιτοντάν. Τώρα για το έλεγχο δύο λεπτά. Κύριε Ματιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές ε, για τις επικοδομητικές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Ε, για τον κύριο από το Frontex. Ε, θα ήθελα να μου πείτε ε, πώς συνεργάζεστε. Είναι ε, μια ενδιαφέρουσα κραποφόρα συνεργασία και ξέρουμε ότι η Κομισιόν μόλις υιοθέτησε μια νέα στρατηγική κατά της εμπορίας ανθρώπων το 2012. Θα θέλαμε να μας πείτε στο επίπεδο αυτό θεωρείτε ότι θα ε, υπάρχουν αποτελέσματα για να καταπολεμηθεί αυτό το τραγικό και πόδινο γεγονός της εμπορίας ανθρώπων, κύριε Αντρέας θα ήθελα να σας πω ότι η παρέμβασή σας ήταν αρκετά συγκεκριμένη και πρακτική, αν μπορώ να πω. Μιλήσατε για σύνδεσμο της εμπορίας ανθρώπων με το οργανωμένο έγκλημα. Σκέφτομαι μια σειρά χωρών όπου θα φαινόταν ότι υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις, σκέφτομαι περίπτωση χάρη τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου ε, επιδεικνύεται να υπάρχει ιδιαίτερο κουράγιο από τις κυβερνήσει, όμως υλοποίησαμε και μια αποστολή στην Καμπότση, παραδείγματο χάρη, και είδαμε πολύ μικρά κορίτσια να εκπορνεύονται ε, και μπροστά στα μάτια όλων και με την ΜΚΟ που βρίσκονται εκεί επί τόπου, εγώ θυμάμαι ότι είδαμε εκεί τους οίκους ενοχής και πραγματικά ήταν τρομερό να βλέπουμε αυτά τα μικρά παιδιά πέντε και εξι ετών, αυτά τα κοριτσάκια να κάνουν το πεζοδρόμιο τη νύχτα και να φεύγουν μαζί με μεγάλους άνδρες και είδαμε μικρά κοριτσάκια που έρχονταν από την Ταϊλάνδη και τις μετακινούσαν στην και τους ε, έκλεγαν και ρωτούσαν τι έκαναν εκεί ήταν πραγματικά τρομερό. Και την επόμενη μέρα μπορώ να σας πω ότι βιώσαμε κάποιες επώδυνες στιγμές, αλλά για αυτά τα κορίτσια ήταν πραγματικά τρομακτικό. την επόμενη φορά, δηλαδή κάναμε, την επόμενη μέρα με συγχωρείτε, κάναμε ένα γύρο με τις ε, ε μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και ε, αυτά τα κορίτσια, τα νάρκο τους έδιναν ναρκωτικά για να μπορέσουν να αντέξουν και οι υπουργοί, οι αρμόδιοι υπουργοί εκεί μας λένε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί πρόκειται για οικογένειες που τελικά πουλούν ένα παιδί για να πουλήσουν τα υπόλοιπα. Εμείς στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν έχουμε το πολιτικό κουράγιο, το πολιτικό θάρρος να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν ξέρουμε ότι το μισό έπ την κατουτζή έρχεται από εμά. Πραγματικά μας λείπει πολιτικό θάρρος. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πέρα από παραδείγματος χάρη να κόψουμε τις προμήθειες των αγαθών. Και πραγματικά σκεφτούμε το παράδειγμα της καμπότση, ε, αλλά Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες για τις οποίες ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να στείλουμε ένα πιο σημαντικό πολιτικό και οικονομικό μήνυμα από αυτό που στέλνουμε σήμερα και πραγματικά συνήθως ε, συνηθίζουμε να γυρίζουμε τη σελίδα, αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μπορείτε να μας δώσετε εσείς ε, κάποια παραδείγματα χωρών όπου πραγματικά υπάρχει πολιτικό θάρρος και υπάρχει τέτοια κατάσταση όπως αυτό που σας ανέφερα. Ευχαριστώ κύριε Ματιά. Σόντερκαρτ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους δύο παρεμβαίνοντας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που μας είπε ο κύριος Βαν Χέλε μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως ε, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την εμπορία των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και μια πτυχή την οποία δεν άκουσα καθόλου. Το θέμα της ζήτησης. Γιατί βεβαίως η ζήτηση είναι αυτή που προκαλεί τα φαινόμενα αυτά. Αυτή οδηγεί την μεταφορά κάποιων ανθρώπων από τη μια χώρα στην άλλη για αυτούς τους σκοπούς. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να ελέγξει ε, την κατάσταση ενημερώνοντας. Δηλαδή αν κανείς δεν ζητούσε αυτήν την ε, εργατική δύναμη με παράνομο τρόπο, δεν θα υπήρχε η οικονομική εκμετάλλευση. Ποιος προκαλεί τη ζήτηση και ποιος ε, έχει οικονομικό συμφέρον και κέρδος από αυτήν την ε, λαθρέα εργασία, παράνομη εργασία. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν πρόκειται πραγματικά για μια εγκληματική δραστηριότητα ή για μια πολύ γνωστή οικονομική δραστηριότητα. Και εδώ θα κάνω μια ερώτηση στην εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Όταν αναφέρεστε σε δουλεία Βεβαίω, τις περισσότερες φορές αναφερόμαστε σε σεξουαλική εκμετάλλευση τη σύγχρονη εποχή. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να σκεφτούμε ποιος προκαλεί αυτή την κατάσταση, ποια είναι η ζήτηση και αν ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας έχει σκεφτεί, έχει προβλέψει κάποια μέσα έτσι ώστε να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση. Όταν παραδείγματος χάρη πάει κάποιος στην Κοπενχάγη σε ένα μεγάλο εργοτάξιο μπορεί να βρει ανθρώπους που εργάζονται με καταναγκαστικό τρόπο. Το ίδιο και στα μεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία. Και εκεί δεν μπορεί να παρέμβει η Frontex. Ποιοι είναι λοιπόν οι τρόποι ε, να αντιδράσουμε εμείς, η κοινωνία των πολιτών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, να εμποδίσουν αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν κάποιες ιδέες και κάποιες προτάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ευχαριστώ κυρία Το Ολοκληρώσαμε τώρα με τους συντονιστές και θα ξεκινήσουμε με τα μέλη. Θα δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά. Την κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πολύ και τους ομιλητές μας εδώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εμπορία ατόμων και για την καταναγκαστική εργασία. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έχουμε την οδηγία, για παράδειγμα, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από τον Απρίλιο του 2013 Έχουμε την στρατηγική που μας παρουσιάσατε και χτες στην Επιτροπή Δικαιοσύνης επίσης ψηφίσαμε για το πακέτο όσον αφορά τα θύματα. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει ακόμα. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε μια περίπτωση που γνωρίζω από την Τσεχία με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί για τα σπαράγγια. Υπάρχουν ε, διάφορα γραφεία τα οποία συνεργάζονται τελικά με μαφιόζικα δίκτυα και προσφέρουν εργαζόμενους για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, με καταναγκαστική όμως εργασία. Οπότε, οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Ποιος λογοδοτεί. Τελικά κανένας δεν διώκεται για τέτοιου είδους εγκλήματα. Η οδηγία μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάνουμε στα εγκληματικά δίκτυα και πώς θα προστατεύουμε τα θύματα. Η ερώτησή μου όμως είναι γιατί φτάνει όπου να είναι ο Απρίλιος του 2013. Δεν ξέρω αν έχει προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία. Πώς όμως μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη κατάσταση και να προλαμβάνουμε τέτοιες ε, καταστάσεις όπως ε, αυτή που διαπιστώσαμε στην ε, Τσεχία. Γιατί τελικά μέσω αυτών των δικτύων τα γραφεία λένε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Και τα θύματα τυχαίνουν, γίνονται βέβαια θύματα εκμετάλλευσης από κάποιους οι οποίοι ποτέ δεν διώκονται. Εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Συνάδελφος Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισαγωγή να πω ότι έχουμε 100 εκατομμύρια γυναίκες ε, που λείπουν από τον ε, πληθυσμό ε, που εξυλοθρεύτηκαν επειδή ήταν γυναίκες και νομίζω ότι ε, είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε γιατί δεν είναι πολιτικά σωστό και μέχρι να το κάνουμε νομίζω ότι θα πρέπει να θέτουμε στο κέντρο το σεβασμό για τις γυναίκες ε, αλλά ε, το ότι κάποιος μετά τη γέννησή του δολοφονείται επειδή είναι κορίτσι είναι πραγματικά τρομερό και αυτό δεν το συμπεριλαμβάνουμε στην ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να το κάνουμε και ήρθε το πληρώμα του χρόνο να το κάνουμε δηλαδή θα έπρεπε ε, ουσιαστικά να λειτουργούμε βάσει του τι είναι δίκαιο και τι είναι όχι, όχι βάσει του πολιτικά ορθού. Και ε, πραγματικά το τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες με τι γυναίκε είναι η λιώψη του ίδιου αλλά αυτή η μεταχείριση των γυναικών κυρίω ε, λαμβάνει χώρα με την ίδια αναλογία σε αυτές τις ε, περιοχές. Η σχέση του οργανωμένου εγκλήματο με την εμπορία ανθρώπων στις χώρες τις οποίες γνωρίζω εγώ καλύτερα ο μεγαλύτερος ε, μεταναστευτικός ε, πληθυσμός ε, δεν μπαίνει καθόλου, δεν επισέρχεται καθόλου στην προσοχή του κοινού. Είναι εκεί, δεν ενοχλούν κανένα, δεν ζητούν κοινωνική πρόνοια, δεν μπαίνουν σε καταλόγους για σπίτια, είναι παράνομοι, τους φέρνουν παράνομα, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι, οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα τους απασχολούν και τους στεγάζουν. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Το πρόβλημα είναι ότι κατόπιν ανήκουν σε αυτού του ανθρώπου που ζουν δουλειά και σπίτι. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι πραγματικό πυρήνα του οργανωμένου εγκλήματο. Δηλαδή, ξεκινά ε, κατά κάποιο τρόπο να πατά το σύστημα, δεν πληρώνει φόρου και ε, κατόπιν ε, φτάνει στο σημείο ένα άνθρωπο να ζητήσει από του ανθρώπου να εργάζονται τζάμπα για αυτού. Διαφορετικά θα του εκθέσει και θα εγκαταλείψουν τη χώρα. Και θέλω να τονίσω τις πόσες δυσκολίες δημιουργεί αυτό και τα προβλήματα που υπάρχουν. Βλέπετε αποδείξεις για αυτό τα θέματα στα κράτη-μέλη. Έχετε κάποια αποδεικτικά στοιχεία από την αστυνομία ή από άλλους φορείς που να εργάζονται με μεταναστευτικές κοινότητες και να ενημερώνουν τους ανθρώπους για, τα μέλη, για τους κινδύνους που διατρέχουν τα ίδια τα μέλη τους. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Βάιλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις ερωτήσεις που έγιναν και στους δύο μιλητές διακρίνουμε πόσα πολλαπλές πτυχές έχει αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία σαν κομμάτια του παζλ. Εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο κομμάτια. Κάποιο ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή ΑΣΕΑΝ και γνωρίζω τι συμβαίνει στι Φιλιππίνε και στην Καμπότζη. Βλέπουμε όμως εδώ μόνο την κορφή του παγόβουνου και σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς θα έπρεπε να οφείσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν ε, κάποιο ρόλο στο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι στην ε, Ταϊλάνδη συνέβη ένα ε, γεγονός, έκλεισαν στη φυλακή κάποιον λόγω σεξουαλικής εκμετάλλευσης ε, παιδιών. Βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πρόστιμα που επιβάλλονται, όμως όταν βλέπουμε οι κυβερνήσεις να καταδικάσουν τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους επιστηρίζουμε και να περάσω στο δεύτερο σημείο, να επανέλθουμε στην Ευρώπη. Η εκπρόσωπος του ΔΟΕ στην αρχή της παρέμβασής της είπε ότι το κύριο πρόβλημα Κοίτα στην ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό διευκολύνει την εμπορία ανθρώπων. Όμως αυτό με ξέπληξε κάπως, γιατί πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κανόνες, έχουμε νόμους, έχουμε εθνική νομοθεσία, έχουμε την Εθνική Νομοθεσία Εργασίας που πρέπει να γίνεται σεβαστή ακόμη και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Υπάρχουν δικαιώματα για αυτούς, υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου, ξεκινώντας από την αστυνομία, τα τελωνία. Και τις αρμόδιες υπηρεσίες ε, για την εφαρμογή της ε, εργατικής νομοθεσίας. Σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι ακριβώ σημαίνει μεμονωμένα σε κάθε κράτο μέλο, όμω σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε να έχουμε εφαρμογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Σταβάρε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, ζητώ συγγνώμη γιατί θα υποχρεωθώ σήμερα να εγκαταλείψω αυτή την Επιτροπή και να πάω στην Υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, γιατί εκεί έχουμε κάποια από τα ζητήματα που συζητάμε. Μ' ακούτε? Έλεγα ότι θα πηγαίνω έρχομαι μεταξύ αυτή τη Επιτροπής και τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί τα θέματα τα οποία συζητούμε ε, ίσω ε, θα έπρεπε να μας οδηγήσουν να κάνουμε μια κοινή συνεδρία των δύο αυτών επιτροπών. Έχω μια-δυο ερωτήσεις για την κυρία Άντρε. Μα ε, είπατε ότι υπάρχουν σήμερα 880.000 θύματα αναγκαστικής, καταναγκαστικής εργασίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Εγώ θα ήθελα να μας παρουσιάσετε κάποια επιμέρους ε, στοιχεία για αυτό το νούμερο. Να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή σε γεωγραφική κατανομή και να μας πείτε και πώς κατανέμεται αυτός ο αριθμός μεταξύ των δύο φίλων. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο συνάδελφος Σόντεργατ σχετικά με τους ε, παράγοντες ε, της ε, παροχής, ε, της ζήτησης ε, από την πλευρά των επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για μεγάλε ή για μικρότερε επιχειρήσει. Πολλέ φορέ επικεντρωνόμαστε σε μικρέ επιχειρήσει, αλλά πολλέ φορέ και μεγάλε επιχειρήσει μπορεί να έχουν ακόμη και 100 εργαζομένου οπού να είναι σε νόμιμο καθεστώ. Εγώ θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή νομοθεσία ύπαρξη, παραδείγματο χάρη, ελάχιστο του μισθού, ανάτομα εργασία. Αν θα μπορούσαν τέτοια μέτρα να αποθαρρύνουν του εργοδότε να ζητούν παράνομη εργασία, εργαζομένου που εργάζονται παράνομα. Γιατί αν θα έπρεπε να πληρώσουν το ίδιο για έναν ντόπιο εργαζόμενο ή για έναν αλλοδαπό εργαζόμενο, τότε δεν θα υπήρχαν πρόσθετα κίνητρα για να προτιμήσουν του παράνομου εργαζομένου. και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με περιπτώσει καταναγκαστική τις εργασίες μεταξύ Ευρωπαίων. Εγώ προέρχομαι από την Πορτογαλία και στη χώρα μου ακούμε κάποιες ειδήσει ότι υπάρχουν Πορτογάλοι εργαζόμενοι που εργάζονται καταναγκαστικά στην Ισπανία ή παραδείγματο χάρη σε χώρε εδώ, στην ευρύτερη περιοχή, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στι κάτω χώρε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν απαντάτε συχνά μια τέτοια πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Συνάδελφος Κοστέλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και για τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Καταρχήν, για τον εκπρόσωπο του Frontex ε, σε σχέση με τη συντονίστρια. Ποια είναι η συντονίστρια που βρίσκεται το γραφείο της και πόσο προσωπικό έχει και ποιους σπόρους. Δεύτερον, σε σχέση με τα θύματα και τη σεξουαλική εκμετάλλευσης, αλλά και της καταναγκαστικής εργασίας. Αλλά ιδίω όταν η συνορική έλεγχη, όταν ο συνορικός έλεγχος η αστυνομία βρίσκει θύματα εμπορίας ανθρώπων, τι διασφαλίσεις δίνεται, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται περισσότερο αν το συλλάβει η αστυνομία και έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες χωρίς χαρτιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα και κάποιες πληροφορίες για το προφίλ των ανθρώπων που είναι αντικείμενο, μάλλον που εμπλέκονται στην εμπορία. Θα με ενδιαφέρε να δούμε την προσωπικότητα ή το πραγματικό προφίλ, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, από πού έρχονται και ποιο είναι το έργο τους στην κοινωνία. Και ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκα στην Ιρλανδία, κυρίω για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευση, Ένα από του τομεί που βρήκα είναι ότι όλη η βιομηχανία διασκέδασης των ελληνικών είναι γεμάτη με ανθρώπου που θα μπορούσαν να είναι θύματα εμπορίας, του βρώμικου χρήματο και διαφθοράς. Και σε πάρα πολλέ χώρε ε, υπάρχει κάποια νομοθεσία που ρυθμίζει αυτό το τομέα, αλλά σε κάποιε χώρε υπάρχουν πολλές μεγάλε διαφορές στην νομοθεσία. Έχετε κάποια άποψη από αυτού και έχετε κάποιε προτάσει ε, για το πώ θα μπορούσαμε να να τον τομέα της ψυχαγωγίας ενηλίκων. Και κάτι άλλο που αναφέρθηκε έχει να κάνει για τη ζήτηση και για παράνομη εργασία και για σεξουαλική εκμετάλλευση. Θα θέλαμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση για σεξουαλική εκμετάλλευση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ε, χωρίς βέβαια να ποινικοποιούμε μάλλον ε, με συγχωρείτε, και με την ποινικοποίηση του ανθρώπου που ζητά, του πελάτη, παρά να ποινικοποιούμε τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και να κατιστούμε πιο δύσκολο για τα άνθρωπα αυτά να έρθουν, να παρουσιαστούν και να καταγγείλουν. Και για την εκπρόσωπο του ΔΟΕ. Συνάντησα πάρα πολλούς μετανάστες που εργάζονται στα σπίτια και παίρνουν το σχάρι μπορεί να κάνουν καταναγκαστική εργασία. Δεν είναι απαραίτητα θύματα ε, εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν προβλήματα με την νομοθεσία όμως. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε από αυτού. Και κάτι ακόμη σε σχέση με το συντονισμό με τις ε, ΜΚΟ, όπως ε, η εκστρατεία ε, σβήστε τα κόκκινα φώτα κτλ. Πώς μπορείτε να συντονίσετε την κατάρτιση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των φορέων που μπορεί να έρχονται σε άμεση επαφή με πολλά από τα θύματα για τα οποία γίνεται λόγος. Ευχαριστώ. Κλείνουμε με τη συνάδελφο Τσαμπόρσκα δύο λεπτά. Τη συνάδελφο Τσαμπόρσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο ομιλητές για την παρουσία τους και για τις προσπάθειες που κάνουν για την καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών ε, δραστηριοτήτων. Πιστεύω πραγματικά ότι το θέμα της προστασίας των θυμάτων, ο εντοπισμός, είναι κάτι που θα πρέπει ιδιαίτερα να μας απασχολήσει. Δεν είναι δυνατόν στους νεώνα που ζούμε να συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, και το ίδιο θα έλεγα βεβαίως και για την σεξουαλική εκμετέλευση, την ε, πορνογραφία, αλλά και την εμπορία οργάνων. Το χειρότερο από όλα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά θύματα που είναι παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να σας ρωτήσω σε τι θέση βάζετε στις προτεραιότητές σας την πρόληψη. Γιατί για να αποφύγουμε να μεγαλώνει ο αριθμός των παιδιών που είναι θύματα αυτής της εκμετάλλευσης, θα ήθελα να μου πείτε τι προληπτική πολιτική, τι προληπτική ε, στρατηγική έχετε για την προστασία των παιδιών. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που κι εγώ άργησα. Δεν θέλω όμως να χάσω αυτή την ευκαιρία τόσο σημαντική για να ρωτήσω αν έχουμε στοιχεία, νούμερα συγκριτικά για τον όγκο χρημάτων που διακινείται μέσω των εγκληματικών αυτών οργανώσεων. Για την εμπορία ατόμων δηλαδή, αν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία ανάμεσα στο διαφυγόν κέρδος από αυτό ή από άλλα πράγματα όπως μπορεί να είναι το εμπόριο όπλων, λαθρεμπόριο νοικοτικών κλπ. Τα άτομα αυτά πώς εντοπίζονται. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είναι οι απαγωγές, αλλά εδώ αυτή η εμπορία με ποιο τρόπο ακριβώς γίνεται. Έπειτα ξέρουμε για τα ναρκωτικά ή για τα όπλα ότι υπάρχει ένα κέρδος όταν ε, τελικά γίνονται κάποιες συλλήψεις ή καταφέρουμε αυτό το διαφυγόν κέρδος να το βρούμε τι γίνεται, πάει πίσω πού, στους φορολογούμενους, στα θύματα, τι γίνεται με αυτό. Και γιατί όγκους μιλάμε, γιατί ποσότητες, γιατί ποσά μιλάμε. Και τα χρήματα αυτά τι γίνονται, αυτόματα μετά πηγαίνουν σε προγράμματα πρόληψης, χρησιμοποιούνται για τα θύματα, πού πάνε. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα να ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να μπορούσαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω το Διευθυντή της Europol που τις προηγούμενες μέρες έστειλε στην Επιτροπή μας μία γραπτή αξιολόγηση για την απειλή που προέρχεται από την εμπορία ανθρώπων και μοιράστηκε από τη γραμματεία την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Η κυρία Ματία αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στην Καμπότζη προλίγου και ε, ακούγοντάς την μου φάνηκε σαν να ξαναείδα όσα είδα σε ένα ντοκιμαντέρ για την εμπορία ανθρώπων στην Καμπότζη και για την εκμετάλλευση αυτών των κοριτσιών που είναι πάρα πολύ μικρά, 4-5 ετών. Εγώ γνώρισα ε, ένα κοριτσάκι που 4 χρονών πολίθηκε από την οικογένειά της ε, για να πάει σε ένα τέτοιο οίκο και κατόπιν κατόρθωσε να το σκάσει και ήταν ε, κλεισμένη στο υπόγειο αυτού του σπιτιού μαζί με ποντίκια και ε, της ε, ξεριζόταν τα μαλλιά γιατί αυτή ήταν να ε, εκπορνευτεί και κατόρθωσε να το σκάσει και ε, μαζί με ένα θείο επειδή πίστευε, πήγε σε ένα θείο της επειδή την πίστευε ότι θα τη βοηθήσει και αυτός την ξαναπούλησε και επειδή αυτό το κοριτσάκι είχε κατορθώσει να το σκάσει έγινε κατά κάποιο τρόπο το σύμβολο των γυναικών αυτών και η κυρία Ματιέ μας δείχνει πως η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών που πηγαίνουν στις χώρες αυτές είναι Ευρωπαίοι. Και πραγματικά πρέπει να υπάρχει το πολιτικό θάρρος να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ε, συμμερίζομαι την αξιολόγησή σας από αυτή τη σκοπιά και κατόπιν η κυρία Γιάννα το τόνισε. Πολύ συχνά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, όταν επικεντρώνουν την προσοχή τους στο έργο αυτής της Επιτροπής, το πρώτο που ε, ρωτούν ε, έχει να κάνει με τις οικονομικές επιπτώσεις, ε, δηλαδή ποιες ε, είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, τι οικονομικά αποτελέσματα έχει μια τέτοια εμπορία, έχετε μια αξιολόγηση τέτοιου είδους. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανχίλ για πέντε λεπτά για να μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με ρωτήσατε για τη διαδρομή από την Νιγηρία. Αεροπορικός, αν έχει χρήματα κανείς και αν μπορεί να πληρώσει για διαβατήρια κτλ. Ορισμένοι που δεν έχουν χρήματα, οδικός και διαθαλάσσεις. Η εκμετάλλευση αρχίζει από την αρχή. Υποσχόμενοι στα θύματα ότι θα βρουν μια καλή δουλειά. Η Μοίρα Φασιλιάδου είναι συντονίστρια που ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών. Τώρα ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πόσο προσωπικό έχει. 6, 7, 8 αλλά κάποιο είναι εδώ από την υπηρεσία της, οπότε ίσως θα μπορούσε να με διορθώσει αν σφάλω. Ασχολείται κυρίως με τον ε, στρατηγικό προσανατολισμό και τον ε, σχεδιασμό στον τομέα αυτό. Υπάρχουν πολλοί φορείς, οπότε χρειάζεται ένας καλός συντονισμός. Εγώ δεν μίλησα για Βέλγους, είπα 400.000 συνοριοφύλακες στην Ευρώπη ολόκληρη. Και δεν είναι μόνο Βέλγοι, είναι από όλες τις εθνικότητες. Μα πάλι μιλήσατε για Βέλγους, δεν καταλαβαίνω. 400.000 συνοριοφύλακες. Βέλγοι που δουλεύουν ως συνοριοφύλακες. Συγγνώμη, δεν σας καταλαβαίνω. Λέω τέσσερα και πέντε μηδενικά μετά. Συνοριοφύλακες. Thousand. Χιλιάδες. Συγγνώμη, Τις μυστικές υπηρεσίες όχι, δεν μπορούμε να τις ε, κυκλοφορήσουμε γιατί τότε και οι εγκληματίε θα τις χρησιμοποιήσουν. Άρα αυτό το χειρίδιο δεν μπορούμε να το μοιράσουμε. Για την Κίνα τώρα για να πάω γρήγορα. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τι γίνεται εκεί. Πρώτα απ' όλα ένας άντρας δεν μπορεί να αποτελέσει θύμα ε, εμπορίας ατόμων, γυναίκες και παιδιά μόνο. Τα νούμερα είναι πολύ πιο ψηλά από αυτά που βλέπουμε εδώ, κυρίως ε, μωρά τα οποία παγάγονται και πολλούνται μετά. Είναι και αυτό μια μεγάλη προτερότητα της κινέζικης κυβέρνησης. Τα ποσά είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ μας. Ε, σίγουρα ε, τα νούμερα είναι πολύ πιο ψηλά από αυτά που έχουμε εμείς τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι οικονομικό το θέμα κυρίως συνήθως, γιατί είναι πολύ ακριβό να συλλέγονται όλοι οι δείκτες και όλες οι πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συλλογή δεδομένων. Γιατί χρειαζόμαστε ε, πολλά δεδομένα για να καταλήξουμε, να συγκεντρώσουμε όλα για μια περίπτωση. Και ε, περνάει ο χρόνος και Φυσικά και υπάρχουν νόμοι που πρέπει να εφαρμόζουν οι χώρες, αλλά δεν γίνεται πολλές φορές. Τα δε δεν κάνουν δηλώσεις τις περισσότερες φορές γιατί φοβούνται ή αλλάζουν τις δηλώσεις τους από φόβο. Στη Γυροπόλη υπάρχουν έτσι και αλλιώς κάποιοι που ασχολούνται με αυτό το θέμα, άρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα γιατί κοστίζει πάρα πολύ ακριβά για την κοινωνία η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Υπάρχει συλλογή δεδομένων, παρόλα αυτά δεν έχουμε αρκετά καλά δεδομένα ή δεν αποφασίζουμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματά μας στη συλλογή δεδομένων. Πρέπει να σταματήσω εδώ και να δώσω το λόγο στην κυρία. Ναι. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικές ε, ερωτήσεις και πολλές. Κοιτάω και την ώρα. Τώρα, όσον αφορά τον ορισμό καταρχήν, ε, εμείς ε, είμαστε πραγματικά ευθυγραμμισμένοι με τους συναδέλφους από τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή το θέμα, αν θέλετε, του εθελοντικού ή όχι, φυσικά και γνωρίζουμε ότι τελικά αυτά τα άτομα είναι θύματα και τελικά απογοητεύονται, διότι άλλα νόμιζαν. Τώρα, τα στοιχεία αυτά κατανέμονται ανατομέα, αναχώρα κτλ. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το κάνουμε. Η ποιότητα των δεδομένων δεν μας το επιτρέπει. Υπάρχουν ε, βεβαίως ε, πολλές χώρες που θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να συσσωρεύσουμε και να κατανείμουμε σωστά αυτά τα στοιχεία. Ε, βοηθήστε μας, ε, με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε με όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, τα χρήματα που προέρχονται από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες εμπορία ανθρώπων. Τα στοιχεία που έχουμε για το 2005 είναι 32 δις και θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή αυτή η είναι πολύ ε, χαμηλά τα ποσά αυτά συνολικά για όλο το χρόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η αριθμή δεν είναι σωστή, μάλλον για 100 δις πρέπει να πρόκειται. Και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε πιο αξιόπιστα στοιχεία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Πολλές ερωτήσεις είχαν αυτό το αντικείμενο. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι καθότι άκουσα από πολλούς από εσάς ότι πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει η ευαισθητοποίηση, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, η ζήτηση, η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες και η ζήτηση για ε, παράνομη εργασία. Τώρα, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το ποιος είναι ο εγκληματίας και αν πρέπει να τιμωρείται ε, το θύμα ή ο θήτης στην περίπτωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παραδείγματο χάρη. Και αυτό δεν το έχουμε ακόμα αποφασίσει. Αλλά το θέμα της ζήτησης και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργοδοσία θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία διαφορετική προσέγγιση ιδιαίτερα όσον αφορά την αλυσίδα της προσφοράς και όταν πρόκειται για παράνομη εργασία, καταναγκαστική εργασία, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εδώ να τιμωρήσουμε και να θεωρήσουμε εγκληματίες όλους τους παρεμένοντες σε αυτή την αλυσίδα. Αυτός που παραδείγματος χάρη που φτιάχνει μπλουζάκια. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, η αναπτυξιακή βοήθεια, πώς μπορούμε δηλαδή να συμπεριλάβουμε θέματα εργασίας και παράνομης καταναγκαστικής εργασίας στις συμφωνίες για την αναπτυξιακή βοήθεια. Το θέμα της μετανάστευσης, του ασύλου επίσης εμπεριέχει τέτοιες πτυχές. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και την ισότητα των φύλων, την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Τώρα, τι μέσα διαθέτουμε, τι εργαλεία χρειαζόμαστε. Όσον αφορά την επιβολή του νόμου, ιδιαίτερα η επιθεώρηση της εργασίας. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει. Έχουμε ξεκινήσει επίσης και μια πιο εξειδικευμένη κατάρτιση για τους επιθεωρητές εργασίες. Υπάρχουν καλές πρακτικές σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα έχουμε εντοπίσει και θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες επιθεωρήσεις. Να εντοπίζονται οι εγκληματίες και βεβαίως να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των επιθεωρητών εργασίας θα πρέπει να συνεργαστούν βεβαίως οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για να προστατεύσουμε τα θύματα κοντά στις κοινότητες των μεθαναστών. Έτσι και αλλιώ οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων είτε δεν υπάρχουν είτε είναι ανεπαρκεί. Και γι' αυτό και ο εντοπισμός είναι πάρα πολύ ελλειπή. Ξέρετε ότι σήμερα τα θύματα φοβούνται, δεν ε, έχουν να κερδίσουν τίποτα από το να καταγγείλουν τους ε, εκμεταλλευτές τους θύτες. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ρωτήσεις. θα απαντήσω αργότερα. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν πολύ συγκεκριμένοι, σεβαστήκατε και το χρόνο και κυρίως σας ευχαριστώ για το ότι παρουσιάσατε αυτές τις στοιχείες από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή μας ε, θα σκεφτεί εις βάθος και θα αναλύσει τα όσα συζητήθηκαν εδώ. Θα ξανασυναντηθούμε γιατί αυτός ήταν ένας πρώτος γύρος ανταλλαγής απόψεων. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ε, συναντήσεις. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα παρά, παράνομη διακίνηση αποβλήτων και άλλες μορφές περιβαλλοντικού εγκλήματος. Ε, αυτά έχουν επίπτωση σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία και πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, είναι χρυσός για τη μαφία αυτή η παράνομη διακίνηση των αποβλήτων και υπάρχει και μια ισχυρή διάσταση διεθνική. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη πτυχή. Θα ακούσαν σήμερα δύο πολύ σημαντικούς ομίλητες που θα μας δώσουν τη δική τους άποψη. Καταρχήν ο κύριος Νιούμαν από ε, την ε, Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Έρευνας με έδρα στο Λονδίνο και ο Σταφέν, ο πρόεδρος της Λαγκαμπιέντε που είναι μία από τις πιο σημαντικέ περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές και από το 79 και κάθε έτος ε, εκπονεί μια έκθεση για την οικομαφία που συντάσσεται με στενή συνεργασία με τις ερευνητικές και δικαστικές αρχές της Ιταλίας. Εγώ είχα την ε, τιμή να παρουσιάσω την έκθεση αυτή την περασμένη εβδομάδα. Είχα κληθεί ως εισηγήτρια και πιστεύω ότι οι ιδέες που θα προκύψουν από αυτή την τελευταία συζήτηση θα είναι πολύ χρήσιμες ε, για τη συνεργασία μας. Την ίδια μέθοδο θα υιοθετήσουμε για τη συζήτηση, 15 λεπτά ο κάθε ομιλητής. Σήμερα όλοι έχουν σεβαστεί το χρόνο τους και εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην ξεπεράσουν τα δύο λεπτά όταν θα πάρουν το λόγο, γιατί διαφορετικά θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε χρόνο από τις απαντήσεις ε, των ομιλητών. Έτσι λοιπόν, 15 λεπτά για τους ομιλητές μας, ε, για τους προσκεκλημένους μας ε, και κατόπιν θα παίρνουν το λόγο πρώτα οι, ο εισηγητής, οι συντονιστές και οι συνάδελφοι για δύο λεπτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με τον κύριο Νιούμαν από τον Οργανισμό Περιβαλλοντικών Ερευνών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η υπηρεσία μου είναι καταστημένη στο Λονδίνο. Είμαστε μια υπηρεσία ερεύνησης εγκλημάτων σε βάρος του περιβάλλοντος. Από το 1984 υπάρχουμε, έχουμε γραφεία στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον και έχουμε και τέρους και στην Ινδία και στην Κίνα και αλλού. Ερευνούμε λοιπόν εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιούμε τις ε, Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις, ε, τα στοιχεία από τις έρευνές μας για να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκλήματα. Υπάρχουν πέντε ειδών είτε πρόκειται για την, το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, είτε πρόκειται για λαθρεμπόριο ουσιών που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος, είτε πρόκειται για παράνομο εμπόριο επικίνδυνων αποβλήτων, είτε πρόκειται για παράνομη ξυλία και εμπορία κλεμμένου ξύλου είτε πρόκειται για την αδήλωτη, παράνομη και άναρχη αλία. Για το, την παράνομη ξυλία υπάρχουν συγκεκριμένες συμβάσεις. Τώρα όσον αφορά το πρώτο, αφορά πολλά είδη. Τίγρη, έχουν μείνει τίγρες που υπάρχουν πολύ λίγες πια. 5.000 δολάρια στην αγορά της Ασίας ε, δικαινούνται για το δέρμα τίγρεων και άλλων ελουροειδών. Όσον αφορά τώρα τις ουσίες που καταστρέφονται στη βάδα του όσοντος, είναι το 20% των θερανθράκων. Η απειλή είναι μεγάλη όσον αφορά το λαθρομπόριο τέτοιων ουσιών. Παράνομη ξυλία τώρα. Στον Αμαζόνιο, στην Ινδονησία, Νοτιοανατολική Ασία. 15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο είναι το κόστος. Υπάρχουν περιφερειακές συμφωνίες και όχι διεθνείς για αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις τώρα των εγκλημάτων αυτών για την αλία και την ξυλία, παράνομη αλία και αξία δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για κλοπή φυσικών πόρων. Έπειτα υπονομεύονται οι κυβερνήσεις, η χρηστή διαχείριση, ενισχύεται η διαφθορά μέσω δωροδοκίας, υπαλλήλων κλπ. Μην ξεχνάμε ότι οι το του θερμοκηπίου έρχονται εξαιτίας της ε, υπερβολικής υλοτομίας, για παράδειγμα. Άρα έχουμε και αλλαγή στο κλίμα. 20% των συνολικών ε, εκπομπών προέρχονται από την απώλεια που έχουμε στα δάση εξαιτίας της παράνομης ε, Πλήττεται και ανθρώπινη υγεία για τα επικίνδυνα απόβλητα, για παράδειγμα όταν ε, αυτά εναποτίθενται εκεί που δεν θα έπρεπε και που στη συνέχεια μολύνεται ο υροφόρος ορίζοντας. Απειλούνται τα οικοσυστήματα και η βιοπικιλία. Και βέβαια το παράνομο εμπόριο υπονομεύει το νόμιμο εμπόριο. τα εγκλήματα αυτά ο κόσμος θα αντιλαμβάνεται σαν να μην αφήνουν πίσω τους θύματα. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή για τον κόσμο όπως είναι τα ναρκωτικά. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό γιατί υπάρχουν πολλά θύματα. Είτε πρόκειται για τη στιβάδα του όζοντος, είτε πρόκειται για άλλες μορφές. Αλλά ακριβώ επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν θύματα, δεν παίρνει την προτεραιότητα αυτό το θέμα. Κι όμως ε, ακόμα και σε χώρες σαν την Ινδονησία, την Βραζιλία, την Καμπότζη υπάρχουν ε, ακτιβιστές υπέρ του περιβάλλοντος που δολοφονούνται. Όμως ο κόσμος δεν δίνει μεγάλη προσοχή. Παρόλο που υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για τις εγκληματικές οργανώσεις. Τα προϊόντα αυτά διακινούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών, διαφορετικών υπήρων και καταλήγουν στην αγορά. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη πρόκληση αντιμετώπιση τέτοιων ε, εγκλημάτων. Θα σας δώσω τώρα κάποια ποσά. Στοιχεία τα οποία πώς να παληθεύσει κανείς, προσπαθώ, είναι στατιστικά δεδομένα που έχουμε για την άγρια ζωή. 7 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Παράνομη ξυλία 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Επικίνδυνα απόβλητα 12 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Παράνομη αλεία 4,2 δισεκατομμύρια και ουσίες που καταστρέφουν το όζον 300 εκατομμύρια δολάρια. Βλέπετε ότι μιλάμε εδώ πέρα για δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα. Πριν από μερικά χρόνια εντοπίσαμε ένα εμπορευματοκιβώτιο που νομίζαμε ότι που διαπιστώσαμε ότι είχε 6 τόνους ελεφαντοστού μέσα. Λαθρεμπόριο δηλαδή. Το οποίο τελικά οδήγησε σε ένα πρόστιμο για τον εισαγωγέα 2.000 δολάρια. Το διασυναριακό έγκλημα. Υπάρχει ένα ξύλο που ονομάζεται Μερμπό από την Παπούα στην Ινδονησία. Ε, πήγαινε στην Κίνα το 2005. 300.000 ε, κυβικά ε, μέτρα το μήνα. Μέσω ενό οργανωμένου δικτύου. Συμμετείχαν ε, σε αυτό κάποιοι αξιωματούχοι από την Παπούα και τη Τζακάρτα, από τη Μαλαισία, τράπεζες οι οποίες πλήρωναν στη Σιγκαπούρη, ε, άλλοι παραγόντες στο Χονγκ Κόγκ, έμποροι από τη Σαγκάη και βέβαια τελικά το ξύλο αυτό το αγοράζανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ας έρθουμε και λίγο στην Ευρώπη. Μίλησα γενικότερα, ας έρθουμε λιγάκι και στην Ευρώπη τώρα και την παράνομη ξυλία εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ παράνομη ξυλία. Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ετοιμάσει μια νομοθεσία που έχει να κάνει με την παράνομη, το παράνομο εμπόριο υλοτομίας και έχει ετοιμάσει και ένα νέο κανονισμό, ο οποίος αρχίζει να ισχύει το 2013. Είναι παράνομο, δηλαδή, να εισάγει κανείς ε, ξύλο που προέρχεται από παράνομη υλοτομία. Ακόμα βέβαια δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Σίγουρα είναι κάτι θετικό, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα τεθεί στην ε, εφαρμογή, γιατί πολλά πράγματα στα χαρτιά είναι μια χαρά, αλλά εφαρμόζονται πολύ πιο δύσκολα. ηλεκτρονικά απόβλητα. Είναι η μορφή αποβλήτων η οποία αυξάνεται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς τελευταία. πολλά, τα κομπιούτερ ή τα άλλα gadgets ηλεκτρονικά, ως απόβλητα τα βρίσκουμε σε διάφορα σημεία. Πρόκειται για 40 εκατομμύρια τόνους τέτοιων αποβλήτων το χρόνο και μόνο το 10% ανακυκλώνεται. Ξέρουμε ότι ε, ορισμένα από αυτά τα απόβλεπτα δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν εκτός Ευρώπης. Όμως γίνεται. Ε, πολλά μηχανήματα ε, διαλύονται στα συστατικά τους και εξάγονται έτσι. Πάνε στην Κίνα, ως επιτοπλίστων. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι. Είναι να ελέγξει τα απόβλητα αυτά. δημιουργώντας ε, δίκτυα και με την ε, οδηγία του 2012. Πέρσι είδαμε ποιος ήταν ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, στα παράνομα αυτά απόβλητα. Πήραμε τηλεοράσει υπολογιστέ, τα διαλύσαμε, τα βάλαμε σε ένα φορτηγό. Τους εφοδιάσαμε ένα tracker για να δούμε ποια είναι η πορεία που ακολουθούν, ποια είναι η διαδρομή η οποία ακολουθούν. Δεν θα έπρεπε να είχαν βγει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν στην Κάνα, στην Άκρα. Και να, που κατέληξαν. Καταλαβαίνετε ότι για το περιβάλλον αλλά και για τους ανθρώπους που επιχειρίζονται αυτά τα υλικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έπειτα έχουμε στην Ευρώπη τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον, χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν ε, απαγορευτεί έτσι ώστε σιγά σιγά να εξαφανιστούν. Το 1997 ένας Γερμανός διαπιστώσαμε ότι σίγαγε 600-700 παράνομα τόνους παράνομα χλωροφθοράνθρακες από την Κίνα. Τότε, χάρη της καλής συνεργασίας του Γερμανού εισαγγελέα με άλλες χώρες, ε, καταφέραμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και να συλληφθεί αυτό ο Γερμανός. Οι χλωροφθοράνθρακες επίσης που πρέπει να εξαφανιστούν έχουν απαγορευτεί από το 2010 και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει εισαγωγή και πώληση. Υπάρχει ζήτηση για αυτές τις χημικές ουσίες. Μία όμως περίπτωση γνωρίζουμε κάτι το οποίο είναι περίεργο. Στην ε, μία κατάσχεση γίνει στην Αμερική που η κατάσταση είναι περίπου ίδια, έχουν υπάρξει πολύ περισσότερες κατασχέσεις. Η Κίνα προσπαθεί να πουλήσει τέτοια χημικά στην Ευρώπη. Πέρυσι, στα σύνορα με τη Ρωσία, υπήρξε άλλη κατάσχεση. Εδώ βλέπετε το δίκτυο αυτών οι οποίοι εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο αυτών των ανακυκλωμένων εντό εισαγωγικών ε, CFCs, κλωροθωροανθράκων καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί αυτό το έγκλημα αν δεν καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς, σας παρουσίασα ε, χοντρικά ποια είναι η κλίμακα του εγκλήματος αυτού. Είναι ένα σοβαρό έγκλημα. Σας έδωσα και κάποια παραδείγματα από την Ευρώπη. Είναι μεγάλη ε, πρόκληση. Τα ποσά αυξάνονταν ελέγξετε 5% των containers, ε, ε, φυσικά θα βρείτε περισσότερα πράγματα, περισσότερες απάτες από ότι αν ελέγξετε το 2%. Άρα χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να μπορούμε να ελέγχουμε περισσότερο. Έπειτα χρειάζεται περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία και πολιτική βούληση. Οι εγκληματίες εύκολα ε, μπορούν να περάσουν τα σύνορα, δυστυχώς. Έπειτα όταν γίνονται κατασχέσεις είτε ελαφαντιστού είτε ουσιών που καταστρέφουν ε, την ε, βάδα του όζοντος, ε, σπάνια καταλήγουν στον εισαγγελέα. Και έπειτα χρειάζεται καλύτερος έλεγχος, μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή πληροφόρηση, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε εκ των προτέρων. Σας είπα ότι από το Ηνωμένο Βασίλειο ηλεκτρονικά απόβλητα κατέληξαν στην Κάνα. Όταν εμείς χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές για να εντοπίζουμε τέτοια εγκλήματα, οι εγκληματίε προχωρούν σε άλλες τεχνικές και ούτω καθεξής. Έχουμε και μερικά καλά παραδείγματα πάντως, γιατί υπάρχουν ειδικευμένε ομάδες για να αντιμετωπίσουν ε, τέτοια περιβαλλοντικά εγκλήματα. Για παράδειγμα, στις κάτω χώρες ή σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε το ΙΜΠΕΛ που είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συνεργάζεται με την Κίνα. Και σιγά σιγά σε διεθνές επίπεδο λαμβάνονται υπόψη πιο σοβαρά τα εγκλήματα αυτά. Είχαμε την δράση Demeter για τα επικίνδυνα απόβλητα. Για να εντοπιστούν δηλαδή πλοία που μεταφέρουν τέτοια απόβλητα. Και η Interpol έχει το δικό της πρόγραμμα με το Eco-Message που είναι ένα πρόγραμμα για ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικά αυτά τα εγκλήματα και γιατί θα έπρεπε να τα λάβετε κι εσείς υπόψη σας. Το Μακάι είναι στα σύνορα Κίνας-Βιετνάμ, βορείως του Ανόη, στην επαρχία Κονγκτσί. Είναι ένα παράδειγμα με πάρα πολλά τέτοια εγκλήματα. 65% κάνουν λαθρεμπόριο μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Νιούμαν. Τώρα θα δώσω το λόγο για 15 λεπτά στον αντιπρόεδρο της Λαγκαμπιέν και τον Στέφανο Σεφάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την πρόσκληση. Με την παρέμβαση αυτή θέλω να σας παρουσιάσω την εμπειρία της οργάνωσής μας και της ομάδας εργασίας που δημιουργήθηκε, που συστήθηκε τα τελευταία στην Ιταλία και μας οδήγησε στο να καταγγείλουμε το φαινόμενο της οικολογικής μαφίας, της οικομαφίας στη χώρα μας. Το 1994 η Λαγκαμπιέντε σύστησε το παρατηρητιό της για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που εδρεύει στη Ρώμη αλλά έχει χίλια κυκλώματα στο τοπικό επίπεδο με συμβούλους και νομικούς. Το 1994 επίσης δημοσιεύτηκε η πρώτη έκθεση για την οικολογική μαφία και κατόπιν ε, τρία έτη αργότερα γίνεται μια ετήσια έκθεση η Λίγκα Βιέντε για να υλοποιήσει την έκθεση αυτή συνεργάζεται με όλες τις διοκτικές αρχές που ασχολούνται με την τήρηση της ε, νομοθεσίας και με ε, τα, ε, τις τοπικές εισαγγελίες και με την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και, εργάζεται και συνεργάζεται και με το Ιταλικό Κοινοβούλιο γιατί από το 1995 υπάρχει μία εξεταστική επιτροπή για την Οικομοφία και για τις παράνομε δραστηριότητε που συνδέονται με αυτό το κύκλωμα. Επίση, συνεργαζόμαστε και με τα τελωνία. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό φορέα ε, για τους ελέγχου ε, στα λιμάνια. Η ομάδα εργασία μεταξύ ε, Ένωσης Πολιτών, δηλαδή πρόκειται για μία μικρόν και μεταξύ αυτών των αρχών καθιστά ένα, καθιστά ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό ως προς τη συνεργασία το 1994 ε, σκεφτήκαμε να εφεύρουμε τον όρο αυτό της οικομαθίας και το 4 χρόνια αργότερα, 5 χρόνια αργότερα μπήκε στο Τζιγκαρέλι, το λεξικό της Ιταλικής γλώσσας ε, και κατόπιν είχαμε έναν ακόμα νεόκοπο όρο, το οικοτέρας, εκομόστρο στα Ιταλικά και θέλαμε ουσιαστικά εκεί να αναφερθούμε στα παράνομα κτίρια αυτό το έργο μας ε, ε, έχει φτάσει σε πολλαπλές εκδόσεις ε, και τον Ιούλιο του 2012 παρουσιάσαμε την τελευταία έκθεσή μας. Είχαμε και συνεργασία και με την εισαγγελία, με είχαμε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και Συνεργαστήκαμε και με τον πρόεδρο του Ιταλικού Κοινοβουλίου που είναι αρμοδίος για την αντιμετώπιση της οικολογικής μαφία και έχουμε μία σύνθεση δεδομένων πέρσι στην Ιταλία. Διεπράχθησαν πάνω από 33.000 αδικήματα, 4 την ώρα δηλαδή το 2011. Είχαμε 305 συλλήψεις, ε, υπήρξαν 28.000 καταγγελίες και είχαμε περίπου 9.000 κατασχέσεις και σε αυτά τα 18 χρόνια εντοπίσαμε 296 ε, φατρίες μαφιόζικες που ασχολούνται με τέτοια περιβαλλοντικά εγκλήματα και επίσης ε, εκτιμήσαμε ε, για το 2011 σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ των κύκλο εργασιών της μαφίας. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε 18 έτη συνεχής εκδόσεις ε, εκθέσεων και το 48% των αδικημάτων ε, συνέβησαν στην ε, τέσσερις περιοχές της Ιταλίας όπου έχουμε μεγαλύτερη παρουσία της μαφίας. Εδώ βλέπετε μια πίτα όπου έχουμε έναν επιμερισμό των περιβαλλοντικών αδειγμάτων που περιγράφουμε στην έκθεση. Πρόκειται για τις παράνομες δραστηριότητες ε, στο τσιμέντο, στις κατασκευές, ε, στα απόβλητα, ε, κατά των ζώων, πυρκαγιές, μπρισμοί. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της οικομοφίας και μιλάμε και για φρεμπόριο επίσης αρχαιοτήτων. Τώρα, παράνομε κατασκευέ, παράνομα κτίρια στην Ιταλία. Το 2011 υλοποιήθηκαν ε, περίπου 26.000 ε, παράνομε κατασκευέ. Στη χώρα μας πρόκειται για ένα τομέα που εγγυάται στην ε, οικομεφία περίπου 2 δισεκατομμύρια έσοδα ετησίως. Βλέπετε οι ιδιοκτικές ε, αρχές έχουν εντοπίσει πάνω από 6.000 αδικήματα. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα. Βλέπετε εδώ ένα λόφο στο Πίτσο Σέλα, στο Παλέρμο στη Σικελία. Εδώ ε, βλέπετε ουσιαστικά ένα σκελετό κτηρίου που υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια περίπου στην ε, Καμπανία σε, ένα, σε μια φανταστική περιοχή. Βρίσκεται στην ακτή. Εδώ βλέπετε μια καταχρηστική τους που έχει ε, χτιστεί στην παραλία και ονομάστηκε ε, ουσιαστικά μάλλον και όσο, όσο καιρό υπάρχει σιγά σιγά ήρθε και η θάλασσα και μπήκε μέσα στη θάλασσα το κτίριο και ε, μιλάμε εδώ για 3.000 ε, παράνομα κτίρια στην ε, Απουλία στο Εθνικό Πάρκο του Γκανκάρνο και βλέπετε ότι καλύπτεται ένα σημαντικό κομμάτι της ακτής της Απουλίας. Άλλα περιβαλλοντικά δικήματα που περιγράφονται στην έκθεση σχετίζονται με το τι συνέβη πέρσι, πρόκειται για τους εμπρισμούς στα δάση, έχουμε αδικήματα κατά της ε, άγριας ζωής, ε, επίσης υπήρχε σημαντική αύξηση των, ε, του λαθρεμπορίου σε σχέση με το 2010, λαθρεμπορίο στα, στα αρχαιολογικά ευρήματα και επίσης είχαμε σχεδόν 14.000 αντικείμενα στον γεωπιστιστικό τομέα οι οργανώσεις ε, της μαφίας ε, διαδραματίζουν και εκεί ένα σημαντικό ρόλο. Τώρα, παράνομος ε, κύκλος διακίνησης των αποβλήπων. Εδώ βλέπετε την παραγωγή ειδικών αποβλήτων στην Ιταλία από το 1997 στο 2007. Σε αυτή την στήλη βλέπετε τις ποσότητες των ειδικών αποβλήτων ε, βιομηχανικής προέλευσης κυρίων που παράγονται, ενώ στη δεύτερη στήλη βλέπετε τα ειδικά αποβλήτα που ε, είναι αντικείμενο διαχείριση σε παράνομες ε, εγκαταστάσεις. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο στυλών είναι η τόνη των ειδικών ε, αποβλήτων που έχουν παραχθεί αλλά δεν έχουν διατεθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εμείς ε, υλοποιήσαμε, ε, συγγνώμη, χρησιμοποιήσαμε αυτή τη στοιχεία και τα μετρήσαμε ουσιαστικά και βλέπουμε ότι κάνουν ένα βουνό ε, σχεδόν 30 εκατομμυρίων τόνων και κάθε χρόνο γεννάται στην Ιταλία ένα νέο βουνό τέτοιων ειδικών αποβλήτων που δεν καταλήγουν σε εγκεκριμένε εγκαταστάσει. Μόνο το 2006 είχαμε το ρεκόρ αυτών των ειδικών αποβλήτων που παρεκτήσαν από δεν κατέληξαν όμω σε νόμιμε εγκαταστάσει. Το 2006 εξαφανίστηκαν στο πουθενά 31 εκατομμύρια δικών αποβλήτων και πράγματι αν ε, τα σκεφτούμε στο χώρο θα καταλάβουν 30.000 τετραγωνικά μέτρα και θα δημιουργούσαν ένα βουνό 3.100 ε, μέτρων, δηλαδή ένα βουνό τόσο ψηλό όσο η Έτνα, το ηφαίστειο έτοιμα στην Ιταλία. Τις ε, δύο τελευταία έτη εμείς ε, είχαμε μια διαφορετική απεικόνηση σε σχέση με τα απόβλητα που παράνομα διακινούνται από την οικολογική μαφία. Αν πάρουμε μόνο τα δεδομένα που γνωρίζουμε, βλέπουμε ότι η βάση των στοιχείων που βασίζονται αντιεκτικές αρχές από το 2010 στο 2010 11 με συγχωρείτε, εξαφανίστηκαν στο πουθενά 2,4 εκατομμύρια ειδικών αποβλήτων. Δεν είχαμε κάποιο πολύ συγκεκριμένο νούμερο που να προέκυψε από τις έρευνες. Μιλάμε για 90. Ε, Μάλλον αυτά τα 2,4 εκατομμύρια φανταστείτε ότι θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μία σειρά 96.000 φορτηγών. Και αν ε, τα αυτά τα φορτηγά στους Ιταλικούς αυτοκινητόδρομους, αν ξεκινούσαμε από την Καλαβρία θα φτάναμε μέχρι το Σαν Μορέτ στην Ελβετία. Πού καταλήγουν τώρα τα ειδικά απόβλητα στη χώρα μας, ε, στην Καπανία, μεταξύ της Νάπολης και της Κατσέρτα. Βλέπετε ε, εδώ ένα χώρο που γεμίζει στη συνέχεια με απόβλητα. Έχουμε εκεί μια παράνομη χαματερή, στη συνέχεια όμως ε, τα θάβουν και δεν φαίνεται πλέον τίποτα, αλλά φυσικά ε, μολύνονται οι υδροφόροι ορίζοντες. Και εδώ βλέπετε και πάλι μια παράνομη χωματερή. Αυτά τα βουνά που βλέπετε δεν είναι βουνά, αλλά πρόκειται για απόβλητα που τα έχουν παράνομα διαθεσική και κατόπιν βλέπετε κάτι ακόμα στην Απουλία. Βλέπετε εδώ σκόνη που προέρχεται από βιομηχανικά απόβλητα από τη Βόρεια Ιταλία. Εδώ βρισκόμαστε στη Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο, είναι γεμάτο από απόβλητα και κατόπιν είμαστε στο Λάτσιο, στο Παλιάνο και αυτές οι μεγάλες σακούλες ε, περιλαμβάνουν απόβλητα που προέρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ βρισκόμαστε στην Καλαβρία, Στο Κροτόνο έχουμε πάλι βουνά από βιομηχανικά απόβλητα που παρήχθησαν τα δεκαετία του 90 από μια κρατική επιχείρηση. Εδώ βλέπετε απόβλητα τα οποία έχουν διατεθεί παράνομα και τα σκορπίζουν ε, στους αγρούς. Εδώ βλέπετε στο Βιτέρμπο, στο Λέτσιο, κάποιες μεγάλες ε, σακούλες που τις έχουν αναποθέσει εκεί. Πρόκειται ε, για απόβλητα από το βορρά. Εδώ πρόκειται για μια καταχρηστική χωματερή, μια τρύπα που έχει γεμίσει με απόβλητα. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η τρύπα. Και στην Ιταλία από το 2001 υπάρχει ένας ε, νέος νόμος για την καταπολέμηση της διακίνησης αποβλήτων. Θεωρήθηκε ε, αδίκημα ως ε, παράνομη δραστηριότητα, παράνομη διακίνηση αποβλήτων, όμως αυτή η νομοθεσία επέτρεψε στις ταλικές αρχές να μπορέσουν να προσφεύγουν σε υποκλοπές, παραδείγματος χάρη, για να ε, παγιδεύουν ε, τους ε, όσους προβαίνουν σε αυτά τα δικήματα, ενώ στο παρελθόν πρόκειτο για πτέσμα, σήμερα θεωρείται πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα αυτό. Και ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποτελεσματικά μέτρα έρευνα και βλέπετε από το 2002 σήμερα χρησιμοποιήθηκαν σε σχεδόν 200 έρευνε που οδήγησαν στη σύλληψη 1200 τέτοιων διακινητών αποβλήτων και ε, ενεπλάκησαν 676 κομπανίες και σε αυτές τις 199 έρευνες 32 αφορούσαν διεθνή διακίνηση που όπου και η χώρα μας και είχαμε να κάνουμε με διεθνή διακίνηση προς 23 ξένες χώρες και οι 10 από αυτές στην Ευρώπη. Μόνο για το 2011, χάρη στη συνεργασία με τα τελωνία, μπορούσαμε να δούμε ότι υπήρχε σημαντική διεθνής διακίνηση από την Ευρώπη προς την Αφρική, τις δεκαετίες του 80 και του 90. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μετακίνηση προς την Ανατολική Οδό και κυρίως προς ε, η Κίνα Ε, στην Κίνα πήγαιναν κάποιες παράνομες εξαγωγές. Εδώ βλέπετε τα υλικά, το πλαστικό καλύπτει σχεδόν ε, το 38% και τα μέταλλα σχεδόν το 48% των ε, αποβλήτων που κατάσχονται και έχουμε δηλαδή αυτά τα δύο υλικά τα οποία είναι αντικείμενο της μεγαλύτερης διακίνησης. Και όπως έλεγα πριν, η Κίνα είναι κυρίως η χώρα τελικού προορισμού βάσει των ερευνών που έγιναν για τις διεθνείς ε, τέτοιε διακινήσεις. Ε, άλλο ο προορισμός είναι το Χονγκ Κόνγκ και άλλες ερεύνες που χρησιμοποίησαν την Ιταλία ως ε, μια τοποθεσία μέσα στο τρίγωνο από τη Ρωσία προς την Ιταλία και μετά στο Χονγκ από το Ισραήλ προς την Ιταλία για να φτάσουν κατόπιν στις κάτω και θα περάσω στα συμπεράσματα. Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση που υλοποιήσαμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία που να μας επιτρέψει να διώξουμε αυτά τα δικήματα και με ποινικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τα προηγούμενα έτη μια οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντο. Η Ιταλία την έχει θέσει εφαρμογή από το 2010 αλλά μάλλον η εφαρμογή δεν είναι και τόσο καλή. Η μεταφορά δηλαδή στο εθνικό δίκαιο δεν είναι και τόσο καλή. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και στη χώρα μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ποινικό δίκαιο, δηλαδή να ενισχύσουμε τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με έλεγχο τέτοιων μετακινήσεων όπως είναι τα τελωνία και να ενισχύσουμε σημαντικές δραστηριότητε που υλοποιούνται από ευρωπαϊκού φορείς όπως Ευρωπόλ, Eurojust και Interpol και τη Unicry. Και κάτι ακόμα που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να πούμε είναι το εξή. Ένα σύστημα για την καταπολέμηση αυτών των παράνομων φαινομένων είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε λεπτομερώς. Για να γνωρίζουμε όμως τις λεπτομέρειες πρέπει να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες όσες μπορούν να προέλθουν από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όλους τους κυβερνητικούς ε, φορείς και την εισαγγελία και τα δικαστήρια και ο καθένας θα μπορούσε να μας δώσει πληροφορίες που αν τις χρησιμοποιήσουμε από κοινού θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα, ένα πλαίσιο συνολικό που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να εγκρίνουμε νέα νομοθεσία, για να αντιμετωπίσουμε νέα φαινόμενα και επίσης να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και νέες έρευνες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα που συνεχώς αναδύονται. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Λαγκαμπιέκτη, τον κύριο Τσαφάνη και θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ. Άκουσα και τις δύο Θα περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Στον ε, κύριο Νιούμαν, σε σχέση με τα περιβαλλοντικά αδικήματα Ε, αναφερθήκατε στην παράνομη αλία. Βρίσκομαι εδώ. Βάσει τη συνεισφορά μας νομίζω ότι θα ήταν καλό να πτύξουμε καλύτερα το θέμα αυτό που πλήθηκε και τη Μεσόγειο. Και έχουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ε, κυρίως ε, που ενελαμβάνονται από την Κίνα, αλλά το θέμα αυτό μπορώ να σα πω ότι αφορά και άλλε περιοχέ. Στον κύριο Τσεφάνη, να θέσω μια άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε κάποιους όρους, οικομαφία, οικολογικό τέρους. Ε, πραγματικά βλέπουμε ότι πλήττεται πραγματικά η επικράτεια. Ε, εσείς μιλήσατε κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, γιατί κάνατε και συγκεκριμένες αναφορές και πολύ σημαντικές ε, σε διεθνή εγκλήματα. Αναφερθήκατε σε κάποια τρίγωνα, σε κάποιες μεταφορές ε, από ένα τομέα σε άλλο και αναφέρεται ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών δικαιωμάτων σε σχέση με την Ιταλία. Βέβαια αυτό το φαινόμενο σίγουρα επαναλαμβάνεται και θα επαναληφθεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Όμως ε, σε σχέση με τις παράνομες κατασκευές, με τα παράνομα κτίρια, τα φθαίρετα, όπως ε, και με τη μαφία στο γεπιστιστικό τομέα. Και αυτό είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ποιο είναι η άποψη μιας ε, τέτοιας ένωσης ε, της δικής ε, σας σε σχέση με τις δυνατότητε που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μιλήσατε για την οδηγία που πρόσφατα μεταφέρθηκε στο ιστορικό δίκαιο από το Εθνικό σας Κοινοβούλιο. Όμως αυτό το χάσμα που υπάρχει τι οδηγεί στην αύξηση των προβλημάτων. Ε, ίσως ε, θα έπρεπε να υπάρχει προσέγγιση των νομοθεσιών ε, μεταξύ των διάφορων κρατών μελών. Μάλιστα, ευχαριστώ. Από το άλλο, ο κύριος Νιούτον um, Ευχαριστώ. Να το μικρόφωνο. Έχω κουραστεί μάλλον. Κύριε Νιούμαν, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση σας. Ποιος σας χρηματοδοτεί, δεν μας είπατε ακριβώς, ε, είστε μη κυβερνητικό οργανισμός, αυτό είναι πολύ γενικό. Δεύτερον, όσον αφορά τους υδροχλωροφεράνθρακες, εγώ ήμουν εισηγητής για μια έκθεση για το θέμα αυτό και πώς μεταφέρονται υπομορφία, αεροζόλ, πώς μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα επικίνδυνα, αυτές οι επικίνδυνες ουσίες. Τρίτο, αυτό το μέρος που μας αναφέρεται στην Κίνα, Μονκάι, κάπως έτσι, πώς γράφεται ακριβώς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε υπέρ ενός ευρωπαϊκού FBI, γιατί προς το παρόν υπάρχει αυτή η συνεργασία, η διασυνοριακή παρόλα αυτά, ε, ποια είναι η λύση σύμφωνα με τη δική σας ε, εμπειρία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κύριε Σαβάνη, σας ευχαριστώ πολύ γιατί μας εξήγησατε πολλά πράγματα. Αυτό που με ξάφνιασε είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα, 92 περιβαλλοντολογικά εγκλήματα συμβαίνουν κάθε μέρα, τουλάχιστον για το περασμένο έτος. Και μόνο 300 συλλήψεις. Φαίνεται ότι στην Ιταλία περνάνε πολύ καλά οι εγκληματίες. Ζωή και κότα. Αυτό που μας είπατε ότι δηλαδή πλέον αντιδράτε. Ποια είναι η αντίδραση των ε, εγκληματικών οργανώσεων, γιατί εδώ μπαίνετε στα χωράφια τους. Όσον αφορά την Κίνα, όσον αφορά τις διακλαδώσεις τους στην Αφρική, τι ακριβώς ζητούν και τι θέλουν να πετύχουν οι Κινέζοι. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία Ματιό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νιώμαν. Μιλήσατε για περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτησή σας. Μας μιλήσατε επίσης και για τα προστατευμένα είδη, ελέφαντες, οι οποίοι συνεχίζουν να, να είναι θύματα των κυνηγών και σήμερα ξέρουμε ότι οι ελέφαντες ουσιαστικά σκοτώνονται για το ελεφαντοστούν. Και είναι ένα πολύ πολύτιμο εμπόρευμα, ιδιαίτερα για κάποιες χώρες όπως ε, στην Κίνα. Υπάρχουν περιοχές εξάλλου που το προϊόν αυτό θεωρείται αφροδισιακό και βεβαίως οι ελέφαντες δεν απειλούνται παντού. Δεν είναι είδο υπό παντού. Σε κάποια μέρη του πλανήτη υπάρχει πληθυσμό ο οποίος ε, πολλαπλασιάζεται με καλούς ρυθμούς. Τι γνωρίζετε για το εμπόριο ακριβώς ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί αυτό το προϊόν. Δεύτερον, κυρία Τσαφώνη, μας δείξατε τρομερές εικόνες και ελπίζω ότι αυτές οι εικόνες, οι οποίες κάνουν πολύ κακό στη χώρα σας, να μην αλλάξουν τόπο για τις ε, καλοκαιρινές τους διακοπές, να έχουν ήδη αγοράσει το εστήριο και να μην μπορούν να τα αλλάξουν και να το ακυρώσουν, γιατί αυτά που μας δείξατε είναι τρομακτικά. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει εγκληματικότητα τέτοιου είδους, όχι μόνο στην Ιταλία και αλλού. Αλλά από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία υπάρχουν ομάδες οι οποίες θέλουν να διαπράξουν αυτού του είδους τα εγκλήματα και την ίδια ώρα εσείς θέλετε να τιμωρήσετε αυτό το έγκλημα, αυτό φάνηκε από την παρουσίασή σας, αλλά μετά την τιμωρία πρέπει να ακολουθήσει καθαρισμός. Τι ε, γνωρίζετε για την κοινωτική χρηματοδότηση όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της μόλυνσης. Για δύο λεπτά, η Γκουε, ο κύριος Σόντεργαρτ. Ε, ευχαριστώ. Δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ε, ε, έγιναν. Κύριε Νιούμαν, μας δώσατε κάποια παραδείγματα, όπως αυτό με έναν πομπό, ο οποίος τοποθετήθηκε στο εσωτερικό αυτών των ε, ε, μηχανημάτων του εξοπλισμού και διαπιστώθηκε η διαδρομή που ακολούθησαν αυτά τα απόβλητα μέχρι την Κάνα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος έχει συμφέρον. Πέρα δηλαδή από τους ενδιάμεσους και το κέρδος που αποκομίζουν, ε, τι άλλο γνωρίζετε για αυτού του είδους το οργανωμένο έγκλημα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ακριβώς πώς ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Κάνα και τι γνωρίζετε για αυτή την παράνομη διακίνηση. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Ο κύριος... Κυρία Μπορσελίνο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, ομιλητές για την εξαντλητική τους παρουσίαση. Θα ήθελα όμως να πω δύο λόγια. Σήμερα το πρωί ακούσαμε την κυρία Αντζελα η οποία μας μίλησε για τις ε, οδούς των ναρκωτικών. Υπάρχει μια ανιχνευσιμότητα, μια δυνατότητα ανίχνευσης ε, της διακίνησης ε, των αποβλήτων. Γιατί αν είναι αλήθεια ότι δυστυχώς ειδήσει που μάλλον τα γεγονότα που μας ανέφερε ο κύριος Κατσάν είναι τραγικά για την Ιταλία. Εμείς ε, στην ε, Ιταλία είναι αλήθεια ότι εμείς ε, δεν βλέπουμε βουνά από απόβλητα, δηλαδή τελικά που καταλήγουν αυτά τα απόβλητα. Υπάρχουν αυτές οι παράνομες χωματερές, αλλά μάλλον είναι περιορισμένες σε σχέση με την ποσότητα ποσότητα, με την ποσότητα των ε, αποβλήτων που διακινούνται. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η Ιταλία απέκτησε αυτή την πολύ σημαντική νομοθεσία. Στις ε, υπόλοιπες όμως ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει τέτοιο αδίκημα. Υπάρχει νομοθεσία που να επιτρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε αυτό το φαινόμενο. Θα ήθελα να κατανοήσω αν ε, η δουλειά που γίνεται από τη Λαγκαμπιέντε στην Ιταλία και γίνεται επίση, υπάρχει πρόθεση να γίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Διαφορετικά θα μείνει ημιτελέ ε, το έργο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά τα απόβλητα, φεύγουν από κάπου, αλλά τελικά δεν μαθαίνουμε ποτέ τι απογίνονται. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Η κυρία Γιάλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, σε αυτή την ροή φαίνεται να υπάρχει ότι έχουμε 23 χώρες και 10 ευρωπαϊκές χώρες αλλά και την Κίνα και τη Ρωσία που λειτουργούν ως ενδιάμεσες. Η Ιταλία δηλαδή θα λειτουργούσε ως ε, μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα. Δηλαδή στην ε, Ιταλία τι συμβαίνει με αυτές τις ροές ε, των αποβλήτων. Τα απόβλητα μετατρέπονται σε κάτι που να μπορεί να μεταφερθεί, να διακινηθεί. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω ποιο ακριβώς ρόλο παίζει η Ιταλία σε αυτή τη ροή. Και στη συνέχεια βρίσκεται αυτά τα απόβλητα, ε, τα κατάσχεται στα τελωνία ή στα λιμάνια ή πηγαίνετε και βρίσκεστε στις παράνομες χωματερές. Και σε σχέση με την παράνομη αλία. Για αυτά που είπε και ο κύριος Γιακολίνο, θέλω και εγώ να ρωτήσω αυτές, ε, αυτά τα κινέζικα σκάφη. Τελικά που δένουν, που αγκυροβολούν στην Νότια Μεσόγειο, στη Μαυριτανία. Υπάρχει και αυτή η θαλάσσια ε, διακίνηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε σε αυτό, θα ήθελα να ξέρω πού εγκυροβολούν. Και για το φαινόμενο που συμβαίνει και στην Ισπανία ε, αυτές τις ε, παράνομες κατασκευές, τα φθαίρετα κτίρια. Τι γίνεται όταν ε, εντοπίζεται αυτά τα κτίρια, στη συνέχεια τι συμβαίνει, δηλαδή στη συνέχεια όταν κάποιος καταδικαστεί πρέπει να καταδευστεί το κτίριο. Και για την, τις πολιτικές αρχές υπάρχει μια νομική βάση που να δίνεται από την νομοθεσία για να παρέμβουν οι αρχές. Και να ρωτήσω επίση ε, τι συμβαίνει με τι καταγγελίε των πολιτών. Υπάρχουν ε, δηλαδή κάποια συστήματα που να μπορεί να πάει ο πολιτή να καταγγείλει και θα έπρεπε να προστατεύονται οι πολίτε αυτοί. Γιατί όταν μιλάμε για μαφία πιστεύω ότι είναι και επικίνδυνη η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει κάποιο τέτοιο οργανωμένο δίκτυο για τι καταγγελίε των πολιτών. Σα ευχαριστούμε για την τελευταία σα παρέμβαση. Γιώτοβα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις ε, ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Θα ήθελα να μου πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τις οργανώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω πρόκειται για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα ήθελα να μου πείτε πώς συνεργάζεστε με τις επίσημες αρχές, με τα δικαστήρια, ε, στις αντίστοιχες χώρες γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αφορά την κοινωνία των πολιτών είναι ότι δεν ε, υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωστοποιηθούν πληροφορίες αυτές. Και μια δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Τσαφάνη. Ακούσαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με τα παράνομα από αυτά την ε, παράνομη διακίνηση αποβλήτων. Αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα ε, προκαλούν, ε, γεννούν, με συγχωρείτε, πάρα πολλά κέρδη για τη μαφία. Συμβαίνει αυτό και στη χώρα μου, στη Βουλγαρία. Μπορείτε να μου πείτε ποια μέτρα παίρνετε για να αναχαιτήσετε αυτή τη διακίνηση και είναι επιτυχή τα μέτρα αυτά. Υπάρχει κάποια γενική ευρωπαϊκή νομοθεσία στην οποία θα μπορούσαμε να βασιστούμε. και υπάρχει και κάποια αντίδραση από τις κυβερνήσεις ε, των αντιστοιχών χωρών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γιώτοβα. Πριν να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση. Αυτό που μας έδειξε ο αντιπρόεδρος Λιγκαμπιέντε σήμερα πραγματικά είναι ένα μέρος ε, της πραγματικότητας. Υπάρχουν ε, ακόμη και πιο ομές, πιο δυνατές εικόνες, αν θέλετε, και θυμόμαστε τι σημαίνει στον Κριτσέντο στην ε, κοιλάδα των ε, ναών. Ε, έχουμε δει πώς γίνεται κάποια κατάχρηση γεών σε ένα βουνό στο Παλέρμο. Είχαμε κάποιες βίλες που είχαν κατασκευαστεί από τον αρχηγό της μαφίας, τον Μικέλε Γκρέκο. Στην έκθεση της Λεγκαμπιέντε αναδύεται το εξής. ότι υπάρχει μια διεθνής διάσταση στο περιβαλλοντικό έγκλημα στην ε, έκθεση που υιοθετήθηκε σχεδόν ομόφωνα τον περασμένο Οκτώβριο, στις 25 Οκτωβρίου, εμείς, ε, χάρη σε αυτή την έγκριση, κατορθώσαμε να δώσουμε την ε, δυνατότητα στο Κοινοβουλίο να εξάγει την θετική του εμπειρία της καταπολέμησης τέτοιου είδους ε, αδικημάτων, γιατί κατόπιν ε, ξεκινά μία σειρά διεθνών αλλά και διευρωπαϊκών ερευνών. Πρόκειται λοιπόν για μία θετική πτυχή επί της οποίας θα έπρεπε να εργαστεί αυτή η υποεπιτροπή. Και Κατόπιν, για την Ιταλία. Στην Ιταλία, η Ιταλία βρίσκεται σε διαδικασία επιπερβάση για το ότι δεν έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μία ευρύτερη αξιολόγηση. Αλλά και η κυρία Μπορσελίνο είπε πού καταλήγουν τελικά αυτά τα απόβλητα. Την περασμένη εβδομάδα εγώ συνάντησα τον επικεφαλής της Καμόρα, τον Φραντσίσκο Μπιντονιέτη και η φατρία του ε, έχει πλουτίσει με αυτή τη διακίνηση αποβλήτων και όταν ε, το ρώτησα αν μπορούσε να με διαφωτίσει με τις ικανότητες που είχε η Καμόρα, μου έδωσε μια απάντηση η οποία μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε πώς όλα αυτά γίνονται χάρη στη διαφθορά και μου είπε πραγματικά να, να ρωτηθείτε άμα ε, εμεί πλουτίσαμε με τα πόβλητα, γιατί και μας τα πόβλητα είναι χρυσός. Ε, αυτό το ρώτησα, με συγχωρείτε, και μου είπε να, ρωτη, να αναρωτηθείτε πώς η Καμόρα μπόρεσε να τα κάνει όλα αυτά. Μπόρεσε να τα κάνει χάρη σε μια διεφθαρμένη πολιτική εν μέρη και επειδή ένα μέρος των θεσμών είναι διεφθαρμένο. Αυτό μας απάντησε λοιπόν. Τώρα λοιπόν να δώσουμε πέντε λεπτά στους κυρίους Νιούμαν και Τσαφάνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την παράνομη αλία, εμείς δεν έχουμε σκάφη, άρα δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην δίωξη αυτού του εγκλήματος. Και βεβαίως εκεί θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αρμόδιους, σε αρμόδιες ομάδες. Όσον αφορά τώρα την οργάνωσή μας, Έχουμε λίγα μέλη, λειτουργούμε με χορηγούς, με χρηματοδότηση εθελοντική και βεβαίως μας χρηματοδοτεί κυρίως ε, αυτή η πηγή, αλλά και έχουμε και μια χρηματοδότηση από, από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση συγγνώμη, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, όσον αφορά την ε, διερεύνηση των εγκλημάτων που σας ε, περιέγραψα. Φυσικά και συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς, με την Ίντερπολ, παραδείγματος για την περίπτωση της Ινδονησίας, παράνομο εμπόριο οξύλιας. Και την τρίτη ερώτησή σας, όσον αφορά το Μονκάι, γράφεται με G, K, A και Y βρίσκεται στα σύνορα Κίνας και Βιετνάμ. Όσον αφορά για τους ελέφαντες, την άλλη ερώτηση. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς σαν αλλά για ιατρικούς σκοπούς ε, το ελεφαντοστούν. Και Κάναμε κάποιες δοκιμές πριν από λίγα χρόνια όσον αφορά την, το νόμιμο εμπόριο ε, στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Και οι πωλήσει αυτής τελικά απλώς κινητοποίησαν την αγορά και πέρσι ήταν η χειρότερη χρονιά η χειρότερη χρονιά και ο όγκος των παράνομων ποσοτήτων που κατασχέθηκαν πολλαπλασιάθηκε. Βεβαίως ε, ξέρετε ότι οι ελέφαντες σε πολλά από τα δάση στην Μοζαμβίκη παραδείγματος χάρη απειλούνται και πιστεύουμε ότι η δίωξή τους ε, καθότι πρόκειται για σπήρες οργανωμένες, ε, οπλισμένες, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει ε, παρά μόνο με την συνεργασία των ε, αρχών και φυσικά βασίζονται σε δίκτυα και κυρίως σε διαφθορά. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί σήμερα να εισάγει νόμιμο λεφαντοστούν από τη στιγμή που δεν έχει διαλευκανθεί και εξαλειφθεί αυτό το εμπόριο. Ήθελα επίσης να σας πω ότι στην ιστοσελίδα μας υπάρχει το System Failure που περιγράφει ακριβώς αυτό που μου ζητήσατε. Επίσης η παράνομη εμπορία αποβλήτων, τα λεγόμενα ε, ηλεκτρονικά απόβλητα και το παράδειγμα που σας έδωσα με το σήμα που μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε Όντως ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, η πληρωμή αν θέλετε είναι και στους ενδιάμεσους αλλά και τελικά και στο σημείο πώληση ε, που ήταν σε αυτή την περίπτωση η Γκάνα. Έτσι είναι επικερδές αυτό το εμπόριο. Ευχαριστώ κύριο Τσεφάνη. Θα ξεκινήσω την ερώτηση του κύριου Γιακολίνου, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά. Η οδηγία η ευρωπαϊκή για την προστασία του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικό μέσο. Ορισμένα συγκεκριμένα δικήματα αφορούν ορισμένες χώρες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή οδηγία, όπως παίρνει το χάρη η κατασκευή αυθαιρέτων κτηρίων, ε, κάτι που το συναντάμε πολύ στη χώρα μας αλλά και σε άλλες μεσογειακές χώρες, δυστυχώς δεν περιγράφεται όπως πρέπει και έχουμε παραδείγματος χάρη και την ε, παράνομη διαχείριση ε, μιας χωματερής και αυτό είναι συγκεκριμένο αδίκημα που συναντούμε σε κάποιες χώρες. Μας, μας ενδιαφέρουν κάποια δικαιώματα που συναντάμε σε κάποιες ζώνες. Στην περιοχή μας όμως δεν υπάρχει επαρκή ορισμός στην Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτών των αδικημάτων. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη να ελέγξει πώς έχει γίνει η μεταφορά της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη και δυστυχώς η Ιταλία το κάνει με λυπή τρόπο. 90 δικήματα την μέρα, μόνο 300 συλλήψεις ε, στην Ιταλία. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι όλα τα περιβαλλοντικά δικήματα στην Ιταλία είναι ε, ουσιαστικά ίσονος ότι ε, είναι τέσματα ή πλημελήματα και ε, μόνο η παράνομη διακίνηση των αποβλήτων θεωρείται κακούργημα στην Ιταλία και μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη όσων τελικά διακινούν τα αποβλήτα αυτά. το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί με όποιον κτίζει ένα παράνομο ξενοδοχείο, ένα αυθαίρετο ξενοδοχείο ή προβαίνει σε άλλα περιβαλλοντικά αντικείμενα που θεωρούνται ίσονο σημασία βάσει τη τελική νομοθεσία. Ε, σίγουρα είναι είναι ανησυχητικέ εικόνε που σα έδειξα. Η Ιταλία είναι ε, πραγματικά εξαιρετική χώρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον τουρισμό στη χώρα μα. Τώρα, ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί για ε, να καταπολεμηθεί η μόλυνση σε κάποια συγκεκριμένα μέρη, σε κάποιες συγκεκριμένες ε, τοποθεσίες ε, και σε τοποθεσίες που έχουν μολυνθεί από τα απόβλητα, έχουν ε, καθυστερήσει οι παρεμβάσεις και μπορώ να σας πω ότι πραγματικά η δράση που αναλαμβάνουμε εκεί δείχνει πόσο πόση μεγάλη κακοδιαχείριση γίνεται ε, στη χώρα μας ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα, πού πηγαίνουν τα παράνομα απόβλητα. Δεν υπάρχει φυσικά μια τέτοια σειρά φορτηγών ε, στα στους δρόμους, ε, πολλές φορές ε, σκορπίζονται στους αχρούς ή άλλες φορές ε, τα ανακατεύουν με τσιμέντο και τα ρίχνουν στα δημόσια έργα. Πραγματικά έχουν βρει πάρα πολλούς τρόπους. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, ή τα ρίχνουν στη θάλασσα. Ναι θα έκλεινα με αυτό, αλλά σας ευχαριστώ για τη βοήθεια, Πρόεδρε. Στο παρελθόν ε, είδαμε γεμάτα πλοία ε, με απόβλητα, κυρίως το κατήριο του 90, τα οποία συνέχεια τα βήθησαν ε, μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα και στις θάλασσες της Ιταλίας το δείγμα τη ε, οργάνωση παράνομη Διακίνηση αποβλήτων ε, που ε, έχει μπει στην νομοθεσία του 2001 δεν το συναντάμε σε άλλα κράτη-μέλη σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως είπε και η Πρόεδρος, θα έπρεπε να το μελετήσουμε λεπτομερώς αυτό το νομοθέτημα, γιατί πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα, πρέπει να ε, αντιγράψουμε και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και για αυτό που είπε η κυρία Μπορσελίνο, αν ε, το έργο της Λιγκαμπιέντα έχει γίνει και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, δεν ε, νομίζουμε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ έδωσα πολύ λεπτομερείς ε, πληροφορίες ε, γιατί το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε στην ε, έκθεση κατά της Μεφίας αποτελεί καρπό με στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τους δικαστές, δηλαδή όλες αυτές οι δυνάμεις δημιούργησαν αυτή τη τόσο παράξενη ομάδα εργασίας μεταξύ μιας ΜΚΟ και των επίσημων θεσμών και καθιστά την Ιταλία μια περίπτωση παραδειγματική, αν μου επιτρέπετε, και θα έπρεπε να ε, ακολουθεί αυτό το παράδειγμα και σε κοινοτικό επίπεδο. Έχουμε μια... Τώρα, αν, αν, το η Ιταλία αποτελεί πλατφόρμα για την παράνομη διακίνηση των αποβλήτων, η Ιταλία χρησιμοποιώντα αυτό το νόμο που ποινικοποιεί ε, τις, ε, οργανώσεις ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, το φαινόμενο αυτό. Εμεί υποψιαζόμαστε ότι παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν χρησιμοποιούν το ίδιο ερευνητικό εργαλείο που και ε, δεν τους επιτρέπει να έχουν μία τόσο ακριβή εικόνα για το τι συμβαίνει, όπως στη χώρα μας παίρνει χάρη. Τώρα τι συμβαίνει με τα φθαίρετα. Ο νόμος λέει κάτι ξεκάθαρο. Οι δήμοι θα έπρεπε να γκρεμίσουν αυτά τα κτίρια, όμως δυστυχώς οι δήμοι δεν ε, κατεδαφίζουν τα κτίρια αυτά τα φέρετα, ακόμη και αν πρόκειται για τόσο κατάφορες περιπτώσεις, όπως ε, αυτό που σας έδειξα πριν ε, στο παλερμο παραδείγματος χάρη, και στο Πίτσιο Σέλα. Και μάλιστα όταν οι κατασκευές έχουν γίνει και από τα κλάν της μαφίας. Τώρα, Αναφέρθηκα στην οργάνωσή μου, είναι μία μική όπου συνεργάζεται με τους θεσμούς, είναι κάτι ιδιαίτερο. Και να κλείσω με την ερώτηση της κυρίας Αλφάνο, εν μέρει απάντησα. το δίκημα, το ότι καθίσταται με παράνομη διακίνηση των αποβλήτων ε, πρέπει να ε, θεσπιστεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να δούμε πώς γινόταν η διαχείριση στο παρελθόν, τα δεκαετία του 90, διαχείριση ορισμένων ειδών ε, αποβλήτων, πολύ επικίνδυνων. Υπήρξε συνεργασία των οργανώσεων της μαφίας με συγκεκριμένα τμήματα του κράτους. Ε, Βλέπαμε παραδείγματος χάρη να βυθίζονται πλοία στη Μεσόγειο. Αυτό αποτελεί ένα σαφές, ένα κατάφορο παράδειγμα για το πώς αυτή η συνεργασία μεταξύ ε, μιας μειοψηφίας που όμως ε, είναι επίσημο τμήμα του κράτους και της μαφίας μας οδήγησαν σε τόσο σοβαρές Περιβαλλοντικέ περιβαλλοντικές καταστροφές. Και μπορώ να σας πω ότι υπήρξε και μία διαστρέβλωση των αποδεικτικών στοιχείων και μία κάλυψη γενικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, στη συνέχεια ε, να γίνει δίωξη των εγκλημάτων αυτών γιατί πραγματικά εξαφάνισαν πάρα πολλές αποδείξεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Λεγκαμπίρτ, ευχαριστούμε και τον κύριο Νιούμαν από την ΙΑΙΑΙ. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, για την παρουσία σας εδώ και σας ευχαριστώ που απαντήσατε. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ άριθμες. Έτσι λοιπόν βλέπετε και πόσο ενδιαφέρεται η Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά και μία παρατήρηση από τον κύριο Νιούτον oh, Όχι, σήκωσα το χέρι μου, δεν ελπίζω να μου δώσω το λόγο, σας ευχαριστώ παρόλα αυτά. Δεν απαντήσατε σε μία από τις ερωτήσεις μου. Τι μπορεί ε, κατά την άποψή σας να κάνει ένα ευρωπαϊκό FBI και την απευθύνω και στους δύο σας. Κοιτάξτε, οποιοδήποτε μηχανισμός που θα βελτιώσει την συνοριακή και υπερεθνική συνεργασία, είτε FBI ή κάτι άλλο, θα μπορούσε να είναι θετικό. Διότι θέλουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων και των κρατών. Η ερώτησή μου είχε να κάνει με τις καταγγελίες των πολιτών. Υπάρχει κάποια στρατηγική που να μπορούν οι πολίτες να καταγγείλουν τέτοια εγκλήματα. Σε ό,τι μας αφορά το Πρατιωτήριο για τα Περιβαλλοντικά Εγκλήματα που ιδρύσαμε το 1994, σκόπευε να γίνει ουσιαστικά και ένας οργανισμός όπου θα γίνονταν οι καταγγελίες από τους ε, πολίτες και ε, η Λαγκαμπίνη ήθελε να παρουσιάζει αυτές τις καταγγελίες στους επίσημους ε, θεσμούς, δηλαδή εν μέρη συνεισφέραμε στο να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στο να καταγγέλουν τα φαινόμενα αυτά. Γίναμε ουσιαστικά για ένας φορέας που δεχόταν αυτέ τι καταγγελίε, τι ε, λάμβανε αυτέ τι καταγγελίε και εμεί τι χρησιμοποιήσαμε αυτέ τι καταγγελίε για να ε, τι συμπεριλάβουμε στην έκθεση εν μέρη και για να τι επισημάνουμε και στι διοικητικέ αρχέ που σε πολλέ περιπτώσει ε, προέβησαν ε, σε κάποιε κατασχέσει ή σε κάποιε παρεμβάσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε και το σημείο αυτό. Ακούσαμε και την τελευταία παρατήρηση της κυρίας Αγιάλα. Στην έκθεσή σας αναφέρεται και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ε, ουσιαστικά ήταν πολιτική αγωγή στη δίκη που καταδίκασε τη μαφία στη Μεσίνα. Υπήρξε λοιπόν και αυτό το είδος αναγνώριση για τη δραστηριότητα της Λεγκαμπιέντε ε, στην ευρύτερη επικράτεια και ουσιαστικά συμμετείχατε και εσείς σε αυτή τη διαδικασία της καταγγελίας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τις συνεισφορές σας. Να συνεχίσουμε τώρα με το τελευταίο πάνελ. Θα ήθελα να καλέσω εδώ τον ε, κύριο Λουίτζι Τσότη, ο οποίος θα μας ε, μιλήσει ε, για, την, ε, για το μετριασμό του κοινωνικού και του οικονομικού αντικτύπου της δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος. Eh. Ευχαριστούμε τον κύριο Λουίτζη Σότη. Η δραστηριότητα της Λίμπερα είναι με δραστηριότητα 360 μοιρών στην Ιταλία και όχι μόνο στη συνεδρίαση των συντονιστών όπου έπρεπε να προτείνουμε τους προσκεκλημένους μας για αυτό το κλάστερ που ασχολείται με την υποστήριξη στα θέματα. Εγώ πρότεινα τον κύριο Τσούτη και υπήρξε ομοφωνία. Έτσι λοιπόν αυτό μας δείχνει πόσο αναγνωρίζεται ο ρόλος της Λίμπερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Η Λίμπερα είναι μια ένωση ε, που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 1995 με στόχο να ζητήσει από την κοινωνία των πολιτών ε, μάλλον να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών να προωθήσει τη δικαιοσύνη. Η κυρία Μπορσελίνο ήταν αντιπρόεδρος της Λίμπερα για πολλά έτη. Εγώ άρχισα να κάνω τα μικρά βήματα στον κόσμο της καταπολέμησης της μαφίας με τη Λίμπερα. Πρόκειται για μια σταθερά λοιπόν σε αυτό τον ε, κόσμο της καταπολέμησης της μαφίας, αλλά πραγματικά πρόκειται για ένα σημείο αναφοράς ε, για τα θύματα και είναι και μια σταθερά ως προς την υποστήριξη σε μια πραγματικότητα που ίσως είναι άγνωστη στην Ευρώπη των μαρτύρων ε, στη δικαιοσύνη. Και όλος αυτός ο χώρος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απάντηση της των πολιτών τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, κύριε Τσότη, έχετε στη σα 20 λεπτά περίπου και κατόπιν θα προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα έχουμε ερωτήσεις ε, από τους συναδέλφους, συντονιστές, εισηγητή και του υπόλοιπους συναδέλφους και κατόπιν θα σας ξαναδώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Καλημέρα σας. Όπως ακούσατε, η Λίμπερα αποτελεί ένα συντονισμό ενώσεων ε, αλλά δεν είναι μόνο κατά της μαφίας, είναι για να οικοδομήσουμε κάποιες διαδρομές δικαιοσύνης και νομιμότητας και αναζήτηση της αλήθειας. Σήμερα στην Ιταλία η Λιμπέρα ε, ουσιαστικά περιλαμβάνει 1.600 ενώσεις μικρές και μεγάλες σε εθνικό επίπεδο που κατόπιν εκπροσωπούνται και σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, αλλά τον Ιούλιο του 2008, εδώ στις Βρυξέλλες, η Λίμπερα ε, δημιούργησε ε, άλλες 120 και έχουμε ε, ουσιαστικά τώρα την οργάνωση Φλερ και θεωρήσαμε ότι οι διαδικασίες που λάμβαναν χώρα στην Ιταλία μας ε, έκαναν να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ε, παρανομίας, της διαφθορές και ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη δική μας χώρα αλλά όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και σήμερα η Φλερ που γεννήθηκε εδώ και εκφράζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη Λίμπερα αλλά και σε διεθνές επίπεδο σήμερα ε, εκπροσωπεί 30 χώρες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και εξετάζει 44 πραγματικότητες. Ε, λοιπόν ε, πρόκειται για ένα δίκτυο που δεν αφορά μόνο την Ιταλική πραγματικότητα, αλλά πρόκειται για ένα δίκτυο που από τη Ρωσία φτάνει μέχρι την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα και υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος. Και ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που μάλλον είναι οι τρεις στόχοι της Λίμπερα. Ο πρώτος στόχος, και πολύ σωστά το υπενθύμησες, είναι η μνήμη. Εμείς έχουμε την ευθύνη της μνήμης ε, να δράσουμε έτσι ώστε η μνήμη να γίνει δέσμευση και κυρίως ε, πρέπει να δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους αυτούς. Ε, συνεχίζουμε να βλέπουμε πάρα πολλούς ε, ορτασμούς ε, ε, ή μάλλον μνημόσυνα, όμως εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε καθημερινή δέσμευση στα θέματα αυτά γιατί είμαστε πεπισμένοι και αυτό το οικοδομήσαμε με τους συγγενείς οι οποίοι έχουν ζήσει στο πετσί τους αυτή τη βία, ότι η μνήμη αφηγείται και αν η μνήμη αφηγείται, το ε, μας βοηθά στο να διαχωρίσουμε το καλό από το κακό και το δίκαιο από το άδικο. Η μνήμη ε, χρησιμοποιείται για να έχουμε ένα, μια νέα κουλτούρα νομιμότητας μέσω της συμμετοχής και εμείς θέλαμε να έχουμε μία ημέρα ε, όπου θα τιμούμε όλα τα θύματα της μαφίας στην Ιταλία. Αυτό το αγγίξαμε σχεδόν. Είχαμε ε, την πρώτη ε, το, ε, το πρώτο μετά ε, το θάνατο του Φαλκόνου ήρθε μια μικροσκοπική κυρία που ήταν ντυμένη με μαύρα ρούχα και είχε και ένα μαύρο μαντήλι στο πρόσωπό της με πήρε από το χέρι και μου λέει πώς δεν λένε ποτέ το όνομα του γιού μου γιατί σήμερα ε, εδώ μνημονεύουμε το θάνατο ε, του δικαστή Βαλκόνε, αλλά ο γιος μου ε, ήταν στο συνοδούς του. Έτσι λοιπόν, οι μητέρες, οι σύζυγοι που έχω χάσει ένα αγαπημένο άτομο, έχουν χάσει ένα άτομο που πέθανε για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας, για τον ίδιο λόγο που πέθαναν και οι άλλοι. Και τουλάχιστον ε, πρέπει να προσδίδουμε την ίδια προσοχή στα άτομα αυτά. Έτσι λοιπόν θέλουμε να έχουμε μία ημέρα το χρόνο όπου στα εργοστάσια, στις πλατείες, ε, στην Ιταλία, στα σχολεία, παντού να υπάρχει μία τέτοια μνήμη. Ήμασταν 200.000 ε, στη Γένοβα φέτος όμως ε, δεν μιλάμε μόνο για τους συγγενείς ε, που συγκεντρώνονται, αλλά συγκεντρώνονται και ένα τμήμα της Ιταλίας, γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο των θυμάτων της μαφίας σε όλη την Ευρώπη με την ίδια δύναμη και με την ίδια αξιοπρέπεια, γιατί όλα αυτά τα άτομα πρέπει ένα-ένα να τα θυμόμαστε στη χώρα μας και ο τρόπος ε, να θυμόμαστε είναι να αναλαμβάνουμε δράση 360 μέρες το χρόνο για να μην έχουμε μόνο ε, εορτασμούς αλλά να υπάρχουν κίνητρα για τη δέσμευση όλων. Έτσι λοιπόν ε, γεννήθηκαν στη χώρα μας κάποιοι σύνδεσμοι, ένας συντονιστικός φορέας στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη για τα θύματα της μαφίας. Και ανακαλύψαμε ότι έτος με το έτος έπρεπε να σκάβουμε για να ανακαλύπτουμε διάφορα ονόματα γιατί δεν υπήρχε κάποιο μητρό που να τα περιλαμβάνει όλα τα ονόματα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο της δέσμευσης και της μνήμης. Τώρα η άλλη μεγάλη διαδρομή για μας, ο δεύτερος μεγάλος στόχος ε, είναι ο πολιτισμός γιατί αυτός αφυπνίζει τις συνειδήσεις. Πρέπει να υπάρχει γνώση και πρέπει να φτάνει κάπως σε όλους. Το, θα το θυμάται και κύριε Μπορσελίνο όταν το 1998 είχαμε εδώ την Επιτροπή της Δικαιοσύνης και υπήρξε ε, μια οδηγία που αφορούσε την καταπολέμηση του εγκληματικότητα και εμείς ήρθαμε για πρώτη φορά εδώ και είχαμε αγωνιστεί για να μην έχουμε μόνο δουλειά σε δικαστικό επίπεδο, σε νομικό επίπεδο, αλλά να υπάρξει και ε, πρόληψη και κατόπιν ε, η οδηγία συμπεριέλαβε και αυτό έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από τα κάτω, από τις ενώσεις, από τις ομάδες, από τα κινήματα. Από εκεί ξεκινάμε και, και θέλουμε να συνεισφέρουμε. Πρόκειται για μια ταπεινή αλλά σημαντική συνεισφορά γιατί προέρχεται από την ιστορία, από την ελπίδα των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν ε, αυτό το θέμα της γνώσης και η διάσταση της εκπαίδευσης είναι αυτή που είναι σημαντική. Έχουμε διαδρομές στα σχολεία, όχι ε, μόνο για να εκπαιδεύσουμε για την ομιμότητα. Πρόκειται για κάτι που αναλαμβάνεται κάθε μέρα, αλλά εμείς ε, μιλάμε για μια αγωγή στην υπευθυνότητα, να είμαστε ενεργοί πολίτες. Ε, πολίτες που αναμειγνύονται, δηλαδή να μιλήσουμε για την υπευθυνότητα της εκπαίδευσης, για να γίνονται σεβαστοί κανόνες. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό βοηθά τους ανθρώπους να οριμάσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί ε, η εκπαίδευση είναι μια μεγάλη διαδρομή στην Ιταλία σήμερα εργαζόμαστε σε 4.200 σχολεία. Δεν πρόκειται για μια μικρή διάσκεψη. Εργαζόμαστε ε, παρέχοντας νέα εργαλεία, καταρτίζουμε τους εκπαιδευτικού. Αλλά για μας το σημαντικό είναι ότι σήμερα 70 σχολές στην Ιταλία έχουν ε, υπογράψει πρωτόκολλα για μάστερ, ε, ορίστε λοιπόν η γνώση, ορίστε ο πολιτισμός, ορίστε ποιες είναι οι διαδρομές για να εμβαθύνουμε περισσότερο και να υιοθετήσουμε αυτή τη μεγάλη πολιτιστική πρόκληση. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην παιδεία που γίνεται από μία κοινωνία ανοιχτή προς το μέλλον, αλλά κάθε πλαίσιο μπορεί να είναι εκπαιδευτικό. Το άλλο μεγάλο στοίχημα, δεν χρειάζεται να το πω σε εσά, αλλά είναι το στοίχημα να στοιχηματίζουμε στους νέους. Μια χώρα που δεν επενδύει στους νέους δεν πιστεύει στον εαυτό της. Όλοι λένε με τα λόγια, εσεί οι νέοι είστε το μέλλον μα, όμως εμεί θέλουμε να είναι οι νέοι το παρόν μας. Γιατί σήμερα βλέπουμε ποιε είναι οι πολιτικές, ε, υποστήριξη στην οικογένεια, αλλά πολλές φορές ε, υπάρχει και απομυθοποίηση του τι συμβαίνει. Γιατί η Λαγκαμπιέντε, παραδείγματο χάρη, που πήρε το λόγο προηγουμένω, αποτελεί τμήμα του ελεύθερου δικτύου και βρίσκεται λοιπόν διάφορε πραγματικότητε με διάφορε ιστορίε, διάφορε διαδρομέ. Και όλοι αυτοί είναι από κοινού, γιατί εμείς είμαστε που κερδίζουμε. Πρέπει να υπάρχουν κινήματα, ομάδες που θα τι βάζουμε μαζί. Και η εμπειρία μας ε, έχει τα ωριά τη, αλλά έχει και τη δύναμή τη πολλοί νέοι συμμετέχουν ε, και μπορούν να υλοποιήσουν και τα, αυτά που τους απασχολούν αν θέλετε, που τους παθιάζουν. Οι νέοι υπάρχουν. Δεν ε, είναι αλήθεια ότι οι νέοι είναι εξαφανισμένοι. Πρέπει όμως να βρουν συγκεκριμένα σημεία αναφορά σήμερα παραποτέ. Και εμείς είδαμε σε πάρα πολλά project ε, που υλοποιήσαμε και που υλοποιούμε είδαμε κάτι τέτοιο. Ο τρίτος μεγάλος στόχος ε, ήταν η κατάσχεση αγαθών από τη μαφία. Υπήρξε ένας νόμος στην Ιταλία που τον ήθελε ο κ. τώρα, ε, έχουν περάσει 30 χρόνια από το θάνατό του. Ένα σικελός ο οποίος γνώριζε τη γη του εις ε, και είχε καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν ε, να υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Και ο Υπουργό Εσωτερικών ε, Ρονιώνη ε, υπέγραψε το νόμο αυτό, όμως τέθηκε σε εφαρμογή μόνο το 1982 στην Ιταλία και λέω μόνο γιατί η Κόσα υπήρχε εδώ και 200 χρόνια, η Καμόρα εδώ και 400 χρόνια υπάρχει στη χώρα μας ε, για να μην αναφερθώ στην ε, Ντράγκεντα στην Καλαβρία. Έτσι λοιπόν μόνο το 1982 έχουμε ε, αυτή την πρόταση νόμου για να θεσπιστεί το αδίκημα αυτό και να μπορούμε να αφαιρούμε τα περιουσιακά στοιχεία των μαφιόζων. Όμως ε, τον σκότωσαν ε, τέσσερις μήνες ε, πριν να ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Σήμερα, μάλλον, συγγνώμη, στη συνέχεια, τέσσερις μήνες μετά δολοφονήθηκε ο Αλμπέρτο Ντελακέζα, τέσσερι μήνε αφού πέρασε η νομοθεσία και ακούστηκαν διάφορε υποσχέσει, δεν θα σα αφήσουμε μόνου, αλλά υπήρξαν και άλλε δολοφονίε και άλλοι θάνατοι. Και μιλάμε για το νόμο που ε, αφορούσε την κατάσχεση. Όμως η κατάσχεση δεν λειτουργήσε και όταν ε, γεννάται αυτό το σύνολο των οργανώσεων εμείς ε, συλλέξαμε ένα εκατομμύριο υπογραφών στην Ιταλία για να ζητήσουμε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο να βελτιώσει το νόμο αυτό, να δώσει συνέχεια στο νόμο αυτό. Όμως... Ε, θέλαμε να χρησιμοποιηθούν και κοινωνικά αυτά τα αγαθά. Θέλαμε να επιστρέψουν ε, στην κοινωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι μιλάμε για μια ηλική αποζημίωση ε, της ζημίας που προκάλεσε η μαφία. Εσείς ε, κατανοείτε ότι αυτό το αγαθό γίνεται πλέον ένα δημόσιο αγαθό και όχι ένα αποκλειστικό αγαθό που τα έχουν στα χέρια τους οι μαφιόζοι. Τώρα κοινωνική χρήση, το κοινοβούλιο ψηφίζει ε, αυτό το νόμο, όμως είχαν συλλεχθεί, όπως σας είπα, ένα εκατομμύριο υπογραφές και τι κάνει η Λίμπερα σε συνεργασία με τους θεσμούς, με τους Δήμους, ε, ζητάοντας από τις κοινότητες να δημιουργήσουν κάποιες συνοπραξίες μεταξύ τους, ο νόμος δίνει αυτά τα αγαθά που έχουν κατασχεθεί στις κοινότητες, στους Δήμους και εμείς προωθούμε ε, κάποιες κοπερατίβες νέων που ε, θέτουν, ε, που χρησιμοποιούν αυτά τα αγαθά. Και εσεί σήμερα στην Ιταλία μπορείτε να πάτε σε ορισμένα καταστήματα, στο υπερκόπ, ε, να αγοράσετε βιολογικά προϊόντα, παραδείγματο χάρη. Και έχουμε τη μοτσαρέλα, το λάδι, τα μακαρόνια. Ο κύριος Απολιτάνο ήθελε την ημέρα που γιορτάζουμε την Ιταλική Δημοκρατία να ε, γιορτάζουμε μόνο με τρόφιμα που έχουν παραχθεί από αυτά τα προϊόντα και προέρχονται από την πραγματική δουλειά της κοπερατίβας ε, η οποία έχει λειτουργήσει ε, με την κατάσχεση των αγαθών αυτών από τους μαφιόζους γιατί στις 2 Ιουνίου ο πρόεδρος είπε αυτά τα αγαθά προέρχονται από αυτά τα εδάφη και διάφορες μαφίες άρχισαν εκείνα τα πάντα. Έβαλαν φωτιά και έκαψαν εκτάρια σε διάφορες περιφέρειες, στο Στράνο, στον Άρο, κοντά στην Κατάνια, στην ε, Απουλία, στο Τορκιαρόλο, στην Καλαβρία. Και υπάρχει λοιπόν η απάντηση των μαφιόζων που θέλουν να πάρουν αυτά τα προϊόντα. Γιατί λοιπόν ε, κάνουν αυτούς τους εμπρισμούς, γιατί θέλουν να σταματήσουν όλη αυτή τη διαδικασία που προσφέρει εργασία σε εκατοντάδες νέους και ε, βλέπουμε ε, αυτά τα προϊόντα στα ράφια και φέρουν το σήμα «Λίμπερα Τέρα, ελεύθερη γη». Όμως ε, μπορεί να ενοχλεί αυτό το σήμα, όμως μας δείχνει ότι είμαστε στον ορθό δρόμο και ε, πρέπει αυτά τα αγαθά και αυτή την κληρονομιά να τη ξαναδώσουμε στο κοινωνικό σύνολο. Και τώρα να αναφερθώ στην οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν Διάφορε ε, διαστάσεις κατά πολέμηση της μαφίας πρόκειται για μια κληρονομιά που πρέπει να ενισχυθεί. Και εμείς από το 1998 συνεργαστήκαμε ε, εδώ με τον Εργόδιο Επίτροπο δικαιοσύνη, ε, έτσι ώστε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει την κατάσχεση και να ψηφίσει μια οδηγία αλλά για να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και ελπίζουμε ότι κατόπιν στο Στρασβούργο θα μπορέσει να εγκριθεί και η κοινωνική χρήση αυτών των αγαθών. Θα πρέπει η συλλογικότητα να χρησιμοποιεί αυτά τα αγαθά. Θα πρέπει να επανέλθουν στη συλλογικότητα τα αγαθά αυτά. Θα πρέπει να ωφελήσουν τόσους νέους. Εμείς ε, αγγίξαμε, ελοπίσαμε αυτό το ε, project, την ελεύθερη γη. Υπάρχουν οι κοπερατίβες και θέλουμε να προωθήσουμε μορφές συνεργασίας ε, για τα αγαθά που έχουν κατασκευθεί. Και είχαμε και προώθηση τουριστική, γιατί ορισμένα ε, από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τον αγροτουρισμό. Και ε, πρόκειται ε, ξέρετε το Κορλαιόνε ήταν ε, αρχηγός της Κοζανόστρα και εκεί αφαιρέθηκαν κάποια περιουσιακά στοιχεία από αυτόν ε, και χρησιμοποιήθηκαν για τον αγροτουρισμό. Όμως το νόημα ήταν ότι μπορούσαμε να το αφαιρέσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να τα ξαναδώσουμε στη συλλογικότητα και να δώσουμε ουσιαστικά δουλειά και αξιοπρέπεια στους νέους. Αυτό ήταν η πιο μεγάλη σφαλιάρα που δόθηκε στη μαφία. Και πρέπει να σας πω ότι μπορούσαμε να δείξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το να ξαναδώσουμε στη συλλογικότητα τα αγαθά αυτά έγινε με τη δέσμευση όλων. Γιατί δεν υπάρχει ένα εγώ, αλλά υπάρχει ένα εμείς. Και μπορούσαμε να δείξουμε ότι ε, μπορούν να συμβαδίζουν οι ηθικοί με την οικονομία. Και σε αυτές τις ε, κατασκευμένα εδάφη καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα και βρίσκουμε, παραδείγματο χάρη, ε, κάποια καταστήματα που φέρουν ε, εκεί ε, το σήμα πρόκειται για τα αγαθά της γεύσης αλλά και της γνώσης και μπορείτε να τα δείτε σε διάφορες πόλεις. Μιλάμε για τη γνώση αλλά και τη γεύση της νομιμότητας, τη Ρέτζιο Καλάμπρια. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός, ε, η παιδεία, το να μπορούμε να δημιουργούμε συγκεκριμένε ευκαιρίε, να δημιουργούνται θέσει εργασία. Βλέπετε λοιπόν πόσο ωφελεί και η μνήμη αλλά και η δικτύωση των συγγενών. Γιατί χρειάζονται λοιπόν στήριξη οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό ήταν το στοιχημά μα, αλλά δεν περιοριστήκαμε εκεί, γιατί έχουμε και ένα ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο δεν ε, μπορούμε να παραμένουμε μόνο θεατές. Ε, πρέπει να υπάρξει συνεργασία για να οικοδομήσουμε από κοινού. Και η μαφία στο ποδόσφαιρο πρέπει ε, να καταγγελθεί. Μάλλον υπήρξε καταγγελία πριν, κάποιους, πριν κάποια χρόνια μέσω ενός βιβλίου. Όμως υπάρχει και δημόσια διαφθορά κύριε και κύριοι, γιατί εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα και τη μαφία. υπάρχουν διάφορες μορφέ νομιμότητα που εξυπηρετούν τη μαφία και έχουμε και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Και πέρσι συλλέξαμε 1.200.000 υπογραφές, τις δώσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και χρειάστηκε να πάμε στα ιστορικά αρχεία του Προεδρικού Μεγάρου. Και ζητήσαμε τι να κάνει η Ιταλία να εφαρμόσει τη σύμβαση του Στρασβούργου του 1999 που θεσπίζει τα δικήματα για τη διαφθορά. Όμως αυτό είναι ντροπή. Γιατί αν δείτε πόσο μικρός είναι ο αριθμός των συλληφθένων, γιατί μιλάμε για 300 άτομα που συνελήφθησαν, αυτό σημαίνει ότι είναι τόσο λίγες συλλήψεις, κάτι δεν λειτουργεί. Χρειαζόμαστε περισσότερους ή λιγότερους νόμους για τη διαφθορά του δημοσίου ε, πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα και έτσι λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε στο σεισμό στην Άκυλα. Η Λίμπερα αμέσω εκπώνησε μια έκθεση με την οποία κατήγγειλε με ονοματιπώνυμα πρόκειτο για ένα φάκελο που το παραδώσαμε. Αμέσως, γιατί η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών είναι υπεύθυνη, είναι παρούσα και έχει κεραίες για να συνεργάζεται χωρίς ρητορική και να συνεισφέρει σοβαρά. Έτσι λοιπόν θεσπίσαμε αυτή την έκθεση για αυτή την αγορά που έγινε μία από τις μεγάλες πηγές εισόδων της μεφίας και η αγορά χρυσού Βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση στη χώρα μας γιατί οι μαφιόζοι ε, χρησιμεύουν ως τράπεζες για να χρηματοδοτούν τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Όμω ε, όλοι μαζί θα νικήσουμε. Ο καθένα συνεισφέρει με τι ικανότητέ του. Ε, δηλαδή, έχουμε διάφορα στοιχεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, ε, τη στήριξη των συγγενών. Όλα αυτά συνεισφέρουν στον να υπάρξει μια αλλαγή. Ανοίξαμε λοιπόν και ένα δίκτυο θηρίδων σε όλη την Ιταλία έναν άξονα δικαιοσύνης για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους να καταγγείλουν. Για να προσφέρουμε και αυτό το χώρο και αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Λουίτσι. Ο κύριος Γεκολίνο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τσότι για την ε, πολύ σαφή του, ιδιαίτερα σαφή του παρέμβαση, ο οποίος ε, μας ανέφερε ορισμένες ε, αρχές που είναι διαπραγμάτευτες, όπως η μνήμη και φυσικά η σχέση με τους επίσημους θεσμούς, το φλερ εκπροσωπείται σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο και είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε τα σημαντικά νομοθετικά παραδείγματα που μας αναφέρετε εσείς, όπως με την κατάσχεση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα της κατάσχεσης και θέλαμε εμείς να εξάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα μοντέλο που είναι επί της ουσίας ιταλικό. Τώρα, σε σχέση με την κατάσχεση έχουμε άριστα μοντέλα, τα οποία εκφράζονται ε, στην έκθεσή σας αλλά και για τους ε, τρόπους της κατάσχεσης σε σχέση με τη χρήση αυτών των εργαθών που κατάσχονται από τη μαφία θα πρέπει και στην Ιταλία να υπάρξει ένας ε, πιο συγκεκριμένη, μια πιο συγκεκριμένη οργάνωση. Θα πρέπει να παρέμβουμε με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καθορίσουμε σε αυτήν ποιος είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι ευθύνε και να καταστήσουμε μια να καταστήσουμε τη χρήση των αγαθών αυτών, αυτών των περιουσιακών στοιχείων απλούστερη αν ε, σε πάνω από 4.000 σχολεία υπάρχει παρέμβαση της Λίμπερα και με πάνω από 70 πανεπιστήμια, αυτό και είναι ένα μοντέλο αριστείας ε, το οποίο θα πρέπει να ε, το εξάγουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν δεν θέλω να κάνω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, απλώς θέλω να καταγράψω αυτή τη δραστηριότητα όλων των οργανώσεων και αυτό αποτελεί μια συγκεκριμένη μαρτυρία για το πώς μπορεί να προωθηθεί η αξία της δικαιοσύνης. Να προσθέσω ότι στην ε, έκθεση έχουμε προβλέψει την προστασία των μαρτύρων ε, και να μπορεί να καταθέσει από απόσταση ο μάρτυρας προκειμένου να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ε, την ε, εξέβριση της αλήθειας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Μποργέτσιο από το ΙΕΦΔΗ. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να αναφερθώ λίγο στο όσα ακούσαμε. Δεν με εξέπληξε το περιεχόμενο, αυτά που άκουσα δηλαδή, Ήμουνα κι εγώ μαζί σας. Είδα από πρώτο χέρι τι έκανε μέχρι τώρα η οργάνωσή σας. Και μάλιστα ο Δον επίσης Συνεπώς θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τις δράσεις αυτές που γίνονται υπέρ των θυμάτων από τα ναρκωτικά. Έτσι, πολλοί νέοι γίνονται πιο παραγωγικοί και δίνουν μια ηθική απάντηση κατά κάποιο τρόπο στην ε, μαφία. Και μάλιστα... αποφεύγοντας μεγάλα κυκλώματα. Θέλω πάντως να υποφεληθώ από τον ε, ομιλητή μας, ο οποίος, ε, ο Ντον Λουίτζι Τσότη, ακούει και παρακολουθεί άτομα τα οποία έχουν συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη κατά το παρελθόν. Έχει μεγάλη εμπειρία. Θέλω όμως να ρωτήσω και κάτι. Πώς γίνεται και πώς θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο για άλλες χώρες, πώς γίνεται η χώρα μας να είχε αστυνομικούς, ανακριτές, ε, δικαστές, οι οποίοι είχαν μια προπτική μακροπρόθεσμα, πώς μετά από αυτή την ε, τόσο ισχυρή πολιτική δέσμευση, μετά από τόσους ανθρώπους που έχουν δουλέψει σε επιτροπές που προσωπικά έχουν αναλάβει τη δέσμευση να κάνουν κάτι τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πώς λοιπόν οι μαφίες αυτές εξακολουθούν να είναι τόσο ισχυρές όπως είναι σήμερα. Πού οφείλεται αυτό, πώς γίνεται. Κροσέτα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω συναντήσει τον Λουίτζι Τσότη και άλλη φορά στις Βρυξέλλες. Είναι συγκινητικό πραγματικά που τον βλέπω. Εγώ ξεκίνησα ως ε, διοικητικός υπάλληλο και με την βοήθεια του Λουίτζι Τσότη και τη Λίμπερα ε, κατάφερα να προστατευτώ από τις απειλές της μαφίας. Όλα αυτά για να σας δείξω τι ρόλο παίζει η Λίμπερα και πώς στηρίζει και τους διοικητικούς. Θυμάσαι τον Νέτα, ο οποίος κατοικούσε 20 χιλιόμετρα από τη Γένοβα και ο οποίος είδε να δολοφονεί το γιος του 16 ετών. Και όταν βρήκαμε το πτώμα, τι έλεγε. Είπε ο γιος μου επέστρεψε. Τον είχε σκοτώσει η μαφία. Καλά κάνεις και θυμίζεις όλα αυτά τα θύματα και τι σημαίνει ο πόλεμος κατά της μαφίας. Υπάρχει και κάτι ακόμα όμως που θέλω να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δώσαμε τη μάχη στην Ιταλία όταν μιλούσαμε για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει ένα σχέδιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν, που θεωρώ όμω ότι δεν είναι πλήρες, είναι ανεπαρκές. Δεν λαμβάνει υπόψη το θέμα των ε, κατασχόμενων αγαθών ή τις κοινωνικές συνέπειες. Θα έπρεπε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε ένα ψήφισμα, να μαζέψουμε υπογραφές από ολόκληρη την Ευρώπη για να δώσουμε τη μάχη μας και σε αυτό το επίπεδο. Βλέπεις δεν είναι δυνατό να επιτρέπουμε μέσω δημοσίων αγορών τελικά η μάφια να παίρνει πάλι πίσω τα περιουσιακά στοιχεία που τους έχουν κατασχεθεί. Η Λίμπερα λοιπόν έχει τον ίδιο ρόλο που είχε και στην αρχή της ιστορίας της. Πρέπει δηλαδή τώρα να δώσει αυτή τη μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω τον Λουίτζι Σότη, με τον οποίο έχω συνεργαστεί για 15 χρόνια στο ιστορικό της Λίμπερα. Η Λίμπερα αποτέλεσε ένα σημαντικό παράδειγμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος γιατί μαζί με εξαιρετικούς αστυνομικούς ε, και μαζί με πολύ προσεκτικούς δικαστές ε, έλειπε κάτι, έλειπε η κοινωνία η οποία έπρεπε με έναν οργανωμένο τρόπο να υλοποιήσει το ρόλο αυτό που δεν μπορούσαν να καλύψουν ε, οι δικαστικοί και οι αστυνομικοί. Ο Παύλο Μπερσελίνο έλεγε ότι η καταπολέμηση της μαφίας δεν μπορεί να γίνει μόνο από τους δικαστές και από τις διοκτικές αρχές, αλλά πρέπει να αποτελεί ένα ηθικό και πολιτιστικό κίνημα που θα, όπου θα συμμετέχουν όλοι. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό το κίνημα μπορώ να το αναγνωρίσω στη Λίμπερα, όχι μόνο γιατί ε, αποτελείται από άτομα που αντιμετώπισαν ε, ισχυρά ε, αυτό το θέμα, αλλά στο παρελθόν δεν υπήρχε ποτέ συντονισμός. Και ακριβώς η Λίμπερα αυτό έκανε, συντόνισε όλα όσοι υπήρχαν στην επικράτεια, αλλά οι άνθρωποι πριν δρούσαν μεμονωμένα. Μιλάμε λοιπόν για την οργάνωση, για το συντονισμό. Νομίζω ότι είναι πάντοτε απαραίτητα και η Λίμπερα αυτά τα έτη μπόρεσε να μας δείξει ότι αυτό ήταν ε, το μέσο, το εργαλείο που έλειπε. Σήμερα στην Ευρώπη ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο και πιστεύω σε αυτά τα τρία έτη έχει γίνει μια σημαντική, ένα σημαντικό έργο και τώρα ε, ξεκινά η κατάρτιση εκθέσεων ή εγγράφων, όπου ίσως και πρώτη φορά αναγράφεται ο όρος μαφία, όπως εμείς αποκαλέσαμε αυτές τις ε, εγκληματικές οργανώσεις. Και θέλαμε να δείξουμε ότι δεν ε, αφορούσε το πρόβλημα αυτό μόνο ε, την Νότια Ευρώπη, την Νότια Ιταλία, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά ίσως και όλο τον κόσμο. Και εγώ νομίζω ότι σήμερα αυτά τα εργαλεία που εντοπίζουμε μέσω της Λίμπερα είναι απαραίτητα και στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει από κοινού ε, να θέσουμε όλους τους πολιτισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτές ήταν οι βελτιστικές πρακτικές ε, που οδήγησαν σε καλά αποτελέσματα στην Ιταλία και μπορούν να αποτελέσουν μια σίγουρη βάση, ένα σημείο αφετηρίας για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε κάποιες ενάρετες διαδρομές, ε, αν θέλετε, όπως έγινε και στη χώρα μας και η παρουσία της ΦΛΕΡ ε, αυτά τα έτη στις Βρυξέλλες Νομίζω ότι ε, ουσιαστικά ε, μας δείχνει ότι ήδη από πριν είχε γίνει κατανοητό ότι αυτό το πρόβλημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε για τη Λιμπερά και πόση προσοχή ε, μας ε, είχαν προσδώσει μέλη του Βουλίου και μας είχαν πει δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης με τέτοια πραγματικότητα. Ίσως γιατί η δραματική κατάσταση που είχαμε εμείς μόλις βιώσει ε, στην Ιταλία και έχει και αντίκτυπο και στη ζωή μας και τις επιλογές μας ίσως δεν υπήρχε αλλού. Έτσι λοιπόν τώρα θα ήθελα να συνεχίσουμε και υπό το φως των εμπειριών της Λίμπερα. Ευχαριστώ. Μήνες Μπεσερίλιο, παρακαλώ. Εσύ, ε, ε, ε, ε Σας ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να εγκαταλείψω αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, κύριο Τσότη και θα ήθελα να σας πω ότι στο Τωρίνο δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μην σας ε, ξέρει και να μην γνωρίζει το έργο σας. Ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε η συνάδελφος Μπορσελίνο όταν είπε ότι στο Κοινοβούλιο πάντοτε μιλούσαμε για εγκληματικές οργανώσεις, αλλά τώρα και χάρη στη δική σας ε, παρουσία, αλλά και στην Προεδρία του κ. Ελφανού και χάρη και κύριο, στους κυρίους ε, Γιακολίνη και Κροτσέτα, πρόκειται για ένα θέμα που προκύπτει συνεχώς. Πάντοτε μιλάμε για τη μαφία και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ θεώρησε ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, γιατί και οι τρει είμαστε θύματα, αλλά εγώ νομίζω ότι τα θύματα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ε, τα θύματα ε, ορούνται θύματα και στη δική μου περίπτωση εγώ είμαι θύμα της τρομοκρατίας, αλλά πρακτικά δεν ε, θα έλεγα ότι είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση, αλλά έχουμε ένα κοινό ιστορικό. Ψηφίσαμε αυτή την οδηγία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία για τα θύματα των εγκλημάτων στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα ελάχιστο πρότυπο, γιατί ξέρω το χάρη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία έχουν πολύ καλή νομοθεσία, για την προστασία των θυμάτων. Ε, φανταζόμαι ότι και η Ιταλία, εσείς θα το γνωρίζετε βέβαια, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπου υπάρχουν πολλά κενά και θα μπορούσαν να υπάρχουν προβλήματα. Τώρα όμως κατορθώσαμε να προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη, να θεωρούνται και οι συγγενείς θύματα και σε πολλές περιπτώσεις ε, όπου δεν υπήρχαν ε, δικαιώματα στα θύματα, έφεση, μετάφραση. Εμείς ε, καταρθέσαμε τώρα να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα και είναι πραγματικό επίτευμα για αυτό το κοινοβούλιο. Ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν για αυτά τα θέματα και για τα θύματα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, θύματα οικογενειακής βίας, θεωρήσαμε ότι έχουν συγκεκριμένες ανακαιότητες, έχουν ιδιαιτερότητες, χωρίς βέβαια να υπάρχει διάκριση από τα άλλα αλλά και ένα θύμα της μαφίας πρέπει να προστατεύεται. Γιατί ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχει και δευτερογενής θυματοποίηση, όπως είχαμε και στην περίπτωση των θυμάτων της τρομοκρατίας. Γιατί αν κάποιο του επιτεθεί, μπορεί να... αυτό σημαίνει ότι θέλει να επιτεθεί σε όλη την κοινωνία. θέλει να τρομοκρατήσουν τους πάντες. Το ίδιο κάνει και η μαφία. Έτσι λοιπόν, απλώ ε, ήθελα να σε ενημερώσω γι' αυτό και να σα πω ότι είμαι στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Ευχαριστώ Τερέσα. Κώστα. Και εγώ. Θα ήθελα να σας ε, πω ότι θρέφω μία πολύ παλιά φιλία ε, με τον κύριο Τσότη για όσα κάνει με τη Λίμπερα και στο πλαίσιο της Φλερ. Και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, γιατί χάρη στη δική τους αποφασιστικότητα αυτή η Επιτροπή μπόρεσε να συσταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα που μας δείχνει πόσο χρειαζόταν ένας χώρος όπου μπορούμε να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε και να γνωρίσουμε και πώς ακριβώς δίνεται αυτή η μάχη σε τελικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω δύο πράγματα. Έχουμε και τον Δαντιέγο, ο οποίος είναι σιερέας, ο οποίος ε, ε, είναι υπεύθυνο ε, σε μια μεγάλη περιοχή της Ρώμης και ε, πραγματικά εργάζονται με τους νέους σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, τους εκπαιδεύουν στην υπευθυνότητα και δεν πρόκειται μόνο για αγωγή στην νομιμότητα, αλλά πρόκειται για μια γενικότερη παιδεία και εγώ νομίζω ότι και στη δική μου Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα να συνεργαστούμε για τα διάφορα προγράμματα που εγκρίνουμε τώρα για τα επόμενα 7 έτη, το Εράσμους, άλλα προγράμματα για την παιδεία, αλλά και για τον πολιτισμό, να βρούμε κάποιες συνέργειες και ευρωπαϊκά δίκτυα πιλωτικά προγράμματα, θα μελετήσουμε όλα αυτά από κοινού, γιατί νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε και να δώσουμε και κάποια συμβολικά μηνύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ με όσα είπε ο κύριο Κροτσέτα που κάλεσε τον ε, κύριο Τσότη να δώσει μια ευρωπαϊκή μάχη για την κοινωνική χρήση των κατασκευέντων περιουσιακών στοιχείων. θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο και είναι σημαντικό να γίνει το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι είναι μια μάχη που πρέπει να γίνει από κοινού, από όλους εμάς και χαίρομαι που το, το, που το αναφέρετε γιατί είναι το κομμάτι που λείπει. Και είναι πολύ σημαντικό, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα όνειρο βέβαια, ε, μπορούμε να έχουμε, έχουμε το σήμα αυτό της ε, Terra Libra, της ελεύθερης θα μπορούσαμε να μιλάμε και για ευρωπαϊκή ελεύθερη γη. Κυρία Γιώτοβα, παρακαλώ. Искам да ви Ευχαριστώ. ευχαριστώ και τον κύριο Τσότη και όλους τους Ιταλούς ε, συναδέρφους, που βέβαια είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις δικές σας δραστηριότητες. Δραστηριότητες οι οποίες όμως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές εκτός Ιταλίας. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί δεν είναι μόνο πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνετε, αλλά και πάρα πολύ χρήσιμα. Και υπάρχει ένα ερώτημα που παραμένει. Πώς προστατεύετε τα θύματα, γιατί η μαφία έχει συνδέσεις με την κυβέρνηση. Κυβέρνηση και μαφία εποφελούνται ο ένας από τον άλλον. Οι δικαστές αντί να τα βάζουν με την ε, μαφία, τελικά τα θύματα είναι αυτά τα οποία διώκονται και τα βάζουν μαζί τους οι δικαστές, επειδή ακριβώς τα θύματα καταπολεμούν τη μαφία. Ευχαριστώ. Πριν να ξαναδώσω στο λόγο στον Τον να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα που φυσικά με αφορά όπως και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ένας από τους στόχους αυτής της Επιτροπής, και το είχαμε πει εξ αρχής, είναι να υπάρξει ένα σχέδιο καταπολέμησης του οργανού κλίματος και αυτό σημαίνει και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ε, των εγκληματιών και χρήση τους για κοινωνικό σκοπό και εμεί ε, θα εργαστούμε προ αυτήν την κατεύθυνση γιατί στην Ιταλία η εμπειρία μας μας έδειξε ότι ο πραγματικό τρόπος για να δώσουμε πραγματικό χαστούκι για να νικήσουμε, για να εξαλείψουμε την ε, δύναμη της μαφίας είναι να τους αφαιρέσουμε τα περιουσιακά στοιχεία. Φαντάζομαι θα εμβαθύνει και ο Δον Λουιτζή, αλλά η κυρία Γετόβα ρώτησε ε, πώς προσφέρετε συγκεκριμένη υποστήριξη στα θύματα. Εγώ θα σας πω ποια είναι η απόψή μου, που νομίζω ότι συμφωνεί και όταν ε, δολοφονήθηκε ο πατέρας μου το 1993, δεν υπήρξε υποστήριξη από τους επίσημους θεσμούς, ε, δεν ήρθε κάποιος πολιτικός να μας υποστήριξει. Ξέρετε, στο σπίτι μας τηλεφώνησε ο Δον Λουίτζι για να μας πει ότι από τη στιγμή εκείνη θα μπορούσαμε να στραφούμε σε αυτούς και ότι θα στεκόνταν δίπλα μας. Προφανώς ε, πρόκειται για μια διαδρομή υποστήριξης, προσέγγισης αλληλεγγύης. Αυτό ζήσαμε εμείς ως θύματα. Κατεκόμη προλίγου αναφερθήκαμε στις μαρτυρίες, στην κατάθεση μαρτύρων. Εγώ πριν ε, τρεις-τέσσερις ημέρες ε, άκουσα τον ε, Υφυπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας επειδή είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις καταθέσεις μαρτύρων. Συχνά Σήμερα το πρωί έκανα μία διαφορά μεταξύ των μαρτύρων και των συνεργατών. Όμως πολύ συχνά στη χώρα μας οι μάρτυρες ε, στέλνουν κάποια ισχυρά μηνύματα, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί πολλές φορές οι δικαστικές αρχές τους ε, επιδικάζουν μία αποζημίωση αλλά η πραγματική αναγκαιότητα για τον μάρτυρα είναι να μπορέσει να επανέλθει στην εργασία του. Γιατί πολύ συχνά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Παίρνει το σχάρι, ένας επιχειρηματίας, αν καταγγείλει κάποια άτομα που έχουν προσπαθήσει να τον εκβιάσουν και να του πάρουν χρήματα και να βγάλουν χρήματα από κάποιον ε, ο οποίος ε, πραγματικά εργάζεται και γίνει τον ιδρώτα του και τελικά καταγγείλει ε, αυτούς τους επικεφαλής της μαφίας, ε, όμως ε, στη συνέχεια όταν ε, προσπαθεί να συμμετέχει στους δημόσιους διαγωνισμούς μπορεί να μην μπορεί να το κάνει και γιατί δεν θα έχει χρήματα, αλλά δεν του δίνουν και αυτούς τους διαγωνισμούς. Κάτι τέτοιο συνέβη στον Πίνο Μορέλη στην Καλαβρία. Και στο Πίνο Μασέρι πριν αρκετά καιρό και είχαμε και άλλον ε, ένα πολύ σημαντικό μάρτυρα, είχαμε την οικογένεια Βερμπάρο, έχουμε πάρα πολλά ονόματα ανθρώπων που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες στη δικαιοσύνη. Ρώτησε κ. Μπουργκέτσε, γιατί δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να νικήσουμε τη μαφία Ίσως γιατί υπάρχουν ε, τόσα πολιτικά κόμματα στην Ιταλία που τελικά συνεργάζονται με τους μαφιόζους ε, ή που υπάρχει ανοχή, ακόμη και το κράτος ε, το κάνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά κοινά συμφέροντα. Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής διακορισμός από τη σκοπιά αυτή. Και κάτι τελευταίο προλίγου, όταν η Τερέσα αναφερθήκε στην εμπειρία της, έγινε λόγο για το εξή όλοι. Θυνόμαστε. αν δεν κάνω λάθος, ε, στις 19 Μαΐου στον Πρίντεση, έγινε μία απόπειρα μπροστά στο σχολείο μορφύλο Φαλκόνε και υπήρξε μία τρομοκρατική επίθεση. Και βρήκε το θάνατο μια κοπέλα. Όμως ε, αυτά τα παιδιά συνεχίζουν ε, να προσπαθούν να επανέλθουν στη ζωή τους, να επιστρέψουν στη ζωή τους. Στην Ιταλία υπάρχει το εξή εγώ κάνω μια πρόταση. Στην Ιταλία υπάρχει ένας νόμος της 3 η Αυγούστου του 2004, ο 206, που προστατεύει τα θέματα της τρομοκρατίας ουσιαστικά προβλέποντας ε, κάποια ωφέλη για αυτούς. Εμείς μπορούμε να ζητήσουμε να μπορούν να υποφεληθούν ε, αυτά τα κορίτσια από αυτό το νόμο γιατί ουσιαστικά εθίγησαν από μια τρομοκρατική πράξη. Ε, αυτά τα παιδιά προσπάθησαν οι άνθρωποι αυτοί να πληγώσουν αυτές τις κοπέλες ε, και κατέστρεψαν για πάντα τη ζωή τους. Λουίτζι, θα σου δώσω κατευθείαν το λόγο για τα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα κύριε Γιακολίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στην Ιταλία έχει σαν βάση ένα νόμο που ψήφισε το Κοινοβούλιο φτιάχνοντας μια εθνική υπηρεσία των κατασκευέντων αγαθών. Δημιουργήθηκαν τη συνέχεια διάφορα συνεταιρισμοί βάλαμε την φαντασία μας να δουλέψει και σήμερα λειτουργούν αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις σε πόρους αρρωγής για να μπορέσουν να ξεκινήσουν. Δηλαδή δεν έχουμε τα εργαλεία για να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους μονάδες. Έπειτα από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατάσχονται, από τα αγαθά τα οποία κατάσχονται, τελικά αυτά πηγαίνουν σε αυτούς τους οργανισμούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που βρίσκουμε εκεί και ναρκωτικά και διάφορα. Ό,τι έχει κατασχεθεί. Η ενισχυτική όμως πληροφορία που έχουμε είναι ότι τα αγαθά τα οποία κατασχέθηκαν από τη μαφία δεν μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν. Και αυτό γιατί έχουν τραπεζική υποθήκη. Και ποιος ε, τη βάζει αυτή την υποθήκη? Ποιος τους ε, επέτρεψε να έχουν αυτή την υποθήκη? 3.000 και λοιπόν ε, ε, περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι τράπεζες θέλουν να τηρηθεί υποθήκη και έχουν δίκαιο στο κάτω-κάτω γιατί και πάλι πρόκειται για χρήματα ε, των πολιτών που δάνεισε τράπεζα. Αλλά από την άλλη λέμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες υποθήκες από τις τράπεζες. Ε, οι τράπεζες λένε εμείς θα πάρουμε τα ακίνητα. Με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Πριν από 15 μέρες ε, υπήρχε η γη του Κρέκοτελ Παπ και η τράπεζα έκανε ένα βήμα πίσω, απέσυρε την υποθήκη και τελικά πάνω στη γη αυτή ελπίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα κονσόρτιουμ για να δημιουργηθεί ένα συνεταιρισμός εργασίας σε δεκάδες εκτάρια γης έτσι ώστε να έχουν αξιοπρεπή δουλειά οι νέοι. Συνεπώς υπάρχουν κάποιες αχτίδες φωτός, αλλά υπάρχουν και αντιφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα δικαιοσύνης ήρθε στην Ιταλία και ήταν και πολύ καλά προετοιμασμένη, μια πολύ συμπαθητική αντιπροσωπεία με την οποία συναντηθήκαμε και θέλησε να δει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί και να δει πώς τα χρησιμοποιούμε. Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Φέτος θα έχουμε λιγότερο λάδι. Γιατί? Γιατί κάηκαν δεκάδες εκτάρια γης. Και μάλιστα να πω ότι η κυβέρνηση ασχολήθηκε αμέσως, έστειλε εγκύκλιο στους νομάρχες και οι μαφιόζοι βέβαια δυστυχώς είναι πιο πονηροί και πιο γρήγοροι. Εκεί όπου υπήρξε έλεγχος στις πυρκαγιές, ξαφνικά έφτασαν 300 πρόβατα. Ξαφνικά, έτσι. Τα οποία ε, έφαγαν το χορτάρι, τα πρόβατα πάνε μια χαρά, οι μαφιόζοι έφεραν προφανώς τα πρόβατα ακριβώς για να φάνε τις καλλιέργειες εκείνους οι οποίες θα δίνανε αξιοπρεπή δουλειά στους νέους που θα συμμετείχαν στις, στους συνεταιρισμούς αυτούς. Υπάρχουν δηλαδή καλά στοιχεία και υπάρχουν και αρνητικά. Η οδηγία αυτή της 12ης Μαρτίου του 2012, κατά τη γνώμη μας, δεν επαρκεί. Χρειάζεται ένα παραπάνω βήμα θα έπρεπε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος του κοινού τα κατασχόμενα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να είναι στα χέρια των μαφιόζων. Είναι δύσκολο. Οι μαφιόζοι τι κάνουνε με τις δραστηριότητές τους. Μας φτωχαίνουν όλους, γιατί μας αφαιρούν κομμάτι της ζωής μας, κομμάτι της περιουσίας μας. Δεν θα έπρεπε λοιπόν τα περιουσιακά του στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τον κόσμο. Κύριε λοιπόν, Μποργέζο, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, η οποία περιλαμβάνει και μέρος της απάντησης για τη δύναμη της μαφίας. Αλλά εδώ δεν θέλω να μιλάω μόνο για την μαφία, γιατί η μαφία σημαίνει πολλά πράγματα. Η δύναμη της μαφίας δεν βρίσκεται μέσα στη μαφία όμως, βρίσκεται εκτός μαφίας. Οι μαφιόζοι αυτά τα άτομα τι δύναμη έχουν, έχουν δύναμη επειδή συμμαχούν με τον επιχειρηματικό κόσμο, με μέλη της κοινωνίας που τους επιτρέπουν να προχωρούν στις διεθνείς τους δραστηριότητες και μερικές φορές έχουν σύνδεση και με την πολιτική. Η δύναμη λοιπόν της μαφίας υπάρχει εξαιτία αυτών των συμμαχιών. Η καταπολέμηση της μαφίας είναι κάτι που προσπαθούμε και το κάνουμε βέβαια και στην κοινωνία, αλλά το κάνουμε και στο κοινοβούλιο. Και πρέπει να γίνει και για την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις. Η καταπολέμηση της μαφίας σημαίνει να έχουν δουλειά οικογένειες, να στηριχτούν, να δώσουμε προτεραιότητα στους νέους, να στηρίξουμε και τις αστυνομικές δυνάμεις και τη δικαιοσύνη που κάνουν ε, αξιοπρόσεχτο έργο. Σήμερα όμως έχουμε μία μαφία η οποία έχει τις ρίζες της στον οικονομικό κόσμο. Είναι δηλαδή μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών έχει γίνει πιο μαφιόζικη γιατί δείχνει ανοχή στη διαφθορά, στην ευνοιοκρατία και στις καταχρήσεις που γίνονται στον οικοδομικό τομέα. Το έχουμε δει αυτό πριν ε, τα ακούσαμε για τα στημένα παιχνίδια, για το τζόγο. Αυτά τα πράγματα είναι που τροφοδοτούν τελικά τη μαφία. Τα τυχερά παιχνίδια. Δέκα δισεκατομμύρια επιτρέπουν στην μαφία να έχει ελεύθερο το πεδίο. Και δεν είναι μόνο στα εγκληματικά παιχνίδια, έχουν ευθύνη και οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν παίρνουν τις σωστές πρωτοβουλίες, δεν ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες. Δεν πρέπει να απλοποιούμε βέβαια, ούτε να γενικεύουμε ποτέ, διότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν θετικό. Πρέπει να δείξουμε θάρρος, να αναλάβουμε δέσμευση. Αύριο θα πάω στην Πόλικα για να θυμηθούμε τον Άντζελο Βασάλο, που και αυτός σκοτώθηκε γιατί δεν λύγησε στις επιθυμίες των μεν και των δε. Κύριε Μπορσελίνο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, πέρα από το ότι σ' αγαπάμε. Είναι ένα αίσθημα που πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία για τα θύματα της τρομοκρατίας. Συμμετείχα σε διάφορες κηδείες θυμάτων της μαφίας. Ο καθένας βάζει το δικό του πετραδάκι που είναι κάτι μικρό, αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε εδώ. Υπάρχει ένα κομμάτι της Ευρώπης που μας παρακολουθεί. Το Μεξικό, να ξέρετε, ζήτησε από τη Λίμπερα να παίξει το ρόλο του, να βοηθήσει τα θύματα με 150 παγωγέ, με 9.000 θύματα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά για το Μεξικό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θύματα από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στο Μεξικό και μας ζήτησαν να βοηθήσουμε τα θύματα έτσι ώστε από τη βάση να φτιαχτεί ένα νέο δίκτυο. Είναι λίγα πράγματα, μικρά, το ξέρω ότι είναι μικρά. Είναι μικρά σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος, αλλά ξέρω επίσης ότι η διαδρομή που γίνεται σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με τα σχολιά. Πολλές φορές έτσι είχαμε σημεία αναφοράς και ακολουθήσαμε πολλές και διαφορετικές διαδρομές. Πρέπει να γίνει μια παραπάνω προσπάθεια, περισσότερο από ποτέ. Ο κύριος Κροσέτα έχει δίκιο, κυρίες και κύριοι. Αυτή η κοινωνική χρήση πρέπει να αποτελέσει πραγματικότητα. Εγώ δεν γνωρίζω όλες τις χώρες που ξέρω ότι στην Ιταλία υπάρχει Λίμπερα. Και εκεί δραστηριοποιείται. Δεν έχω χρόνο μπροστά μου για να σας πω πολλά ακόμα. Θέλω απλώς να σας ε, πω τέσσερα πραγματάκια ακόμα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή κάποιος κατάλαβε ότι κάτι αλλάζει στη ζωή μας. Χρειάζεται πολύ ταπεινοφροσύνη, χρειάζεται συνέχεια και χρειάζεται βούληση να προχωρήσουμε στις πολιτικές μας ε, μαζί και να υπάρξει ευθύνη από όλου. Οι πολιτικοί έχουν τη δικιά τους την ευθύνη, εμείς οι πολίτες έχουμε τη δικιά μας την ευθύνη. Διαφορετική ρόλη, αλλά αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας με αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Δον ευχαριστώ και τους διερμηνείς για τον παραπάνω χρόνο. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 9 με το πρωινό πάνελ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.